Good morning. Uh, Καλημέρα. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει διαδίκτυο, δηλαδή στο δίκτυο του Κοινοβουλίου, αλλά δεν το χρειάζεστε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, σήμερα και ολόκληρο το πρωινό θα εξετάσουμε τα διάφορα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία ασφάλεια τροφίμων και αυτό είναι μέρος ε, της ημερήσιας διάταξής μας. Εμείς λοιπόν θα επικεντρωθούμε στα τρία που έχουν να κάνουν με το κλίμα, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Έχουμε τρεις εμπειρογνώμονες εξωτερικούς που έχουν εκπονήσει μελέτες για το τι μπορούμε να περιμένουμε για τα διάφορα αυτά θέματα θα μας ε, παρουσιάσουν τις, ε, τις εργασίες τους αυτές. 10 λεπτό καθένας και πριν τις 12.30 θα πρέπει να έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, μετά από κάθε παρουσίαση θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Οι τρεις εμπειρογνώμονες που έχουμε μαζί μας σήμερα και μας είπαν ότι να ξέρετε ότι επειδή είναι ευρύ το θέμα, έχουμε ζητήσει την άποψη κι άλλων, γιατί δεν είναι εμπειρογνώμονε σε όλες τις λεπτομέρειες όλων των επιμέρους ε, θεμάτων που θα εξετάσουμε σήμερα, αλλά θα μας δώσουν μια γενική επισκόπηση και μετά θα μπορέσουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας. Οι τρεις που έχουμε είναι πρώτα Ιάν και Χέρολτ από το ΕΚΟ Ινστιτούτο που θα μας μιλήσει για την κλιματική αλλαγή. Έχουμε τη Φρασίσκα Βόλφ που είναι επίσης από το ίδιο Ινστιτούτο ΕΚΟ που θα μας μιλήσει για τις περιβαλλοντικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά έχουμε τον Νίκολα Πουσκαρεφ από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία που θα μας μιλήσει για την υγεία. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα περάσουμε στο πρώτο θέμα που είναι η κλιματική αλλαγή, πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, κατάσταση πραγμάτων σήμερα και ποιες είναι οι μελλοντικέ προκλήσεις. Θα δώσω το λόγο στην Άνκε Χέρολτ, λοιπόν για να μας παρουσιάσει τι να περιμένουμε. 15 λεπτά, 15 λεπτά έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Μα ζητήθηκε στη μελέτη να εξετάσουμε την τρέχουσα νομοθεσία. Πρώτα απ' όλα ποιοι είναι η σημερινοί στόχοι και ποια είναι η σημερινή στρατηγική. Και μετά να δούμε τις μελλοντικές προκλήσεις. αρθρώσαμε λοιπόν τις μελλοντικές προκλήσεις στους τομείς που έχει ήδη αναφέρει και προωθεί η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φόντερ Λάιεν, ώστε να δούμε τι θα γίνει στην επόμενη θητεία. Και κοιτάμε και ποια είναι και τα κενά και αδυναμίες στην εφαρμογή της πολιτικής περιβάλλοντος. Δεν φαίνεται καλά η διαφάνεια, αλλά θα προσπαθήσω να εξηγήσω ποιες είναι οι τάσεις των αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, θα σας το εξηγήσω. Για το 2020, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μείον 20% σε σχέση με το 1990. Και μετά για το 2030 είναι μείον 40% σε σχέση με το 1990. Και αυτός είναι ο στόχος που έχει υποβάλει στη Συμφωνία των Παρισίων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον μείον 40%. Μακροπρόθεσμα τώρα, για μέχρι το 2040, δεν έχουν ακόμα καθοριστεί οι συντελεστές στην νομοθεσία, αλλά υπάρχει η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει για το 2050 μείον 80 με μείον 95% εκπομπές. Το μαύρο κομμάτι που βλέπετε εδώ είναι οι σημερινές εκπομπές και βλέπετε ότι ήδη έχουμε Είμαστε λίγο πιο κάτω από το στόχο του 2020 και μετά είναι διακεκομένες οι πράσινοι και οι πορτοκαλί που δείχνουν προβλέψεις για το μέλλον. Και βλέπετε ότι είναι λίγο πάνω ακόμα από τους στόχους του 2030. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται επιπλέον προσπάθεια, επιπλέον μέτρα για να πετύχουμε τον στόχο του 2030. Θα επανέλθω σε αυτό όμως αργότερα. Τώρα, σε σχέση Συνολικά με τους στόχους για το περιβάλλον υπάρχουν διάφορες ε, προκλήσεις. Σύμφωνα με τις ε, συμφωνίες των Παρισίων, του χρόνου θα υπάρξει μια αναθεώρηση των εθνικά καθορισμένων ε, εισφορών. Οπότε θέλουμε κάποια ενημέρωση της συμφωνίας των Παρισίων. Γίνεται συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα για το κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε πιο φιλόδοξους στόχους για το 2030. Στην πρόταση της κυρίας Φοντερ Λάιεν αναφέρεται ότι θα ήθελε να πάμε προς το μείον 50%. Και αν και οι άλλες οικονομίες δείξουν υψηλότερες φιλοδοξίες, θα μπορούσαμε να πάμε και στο μείον 55% μείωση των εκπομπών σε σχέση πάντα με το 1990. Και αυτό αναφέρεται και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της προηγούμενης θητείας που στηρίζει ε, πιο φιλόδοξους στόχους. Στη συνέχεια ε, συζητάμε και για τους μακροπρόθεσμους στόχους, για το 2050 δηλαδή, να πετύχουμε την ουδετερότητα όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα. Μείον 80 με μείον 95% λέμε τώρα και είναι κάτι που έχει ήδη συζητηθεί στο Συμβούλιο και το στήριξαν πολλές χώρες μέλη, όμως υπάρχουν και κάποιες που αντιτίθενται. Θα είναι πάντως στην εμερήσια διάταξη της Φιλανδικής Προεδρίας και πάλι. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει αλλαγή και στην νομοθεσία όσον αφορά ε, την κλιματική αλλαγή, προκειμένου να τεθούν στην νομοθεσία οι στόχοι του 2005 και να καλυφθεί έτσι η περίοδος 2020 με 2050. Μια άλλη πρόταση είναι ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα μεταξύ περιφερειών, τοπικών κοινωνιών, κοινωνίας των πολιτών και σχολείων. Ένα σημαντικό σημείο για να στηριχθεί η πολιτική αυτή είναι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021 μέχρι 2017 θα έπρεπε να λέει 2027. Αυτό είναι το σωστό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αύξηση των δαπανών ε, υπέρ του κλίματος από 20% σε 25%, κάτι το οποίο αντιστοιχεί σε 320 δισεκατομμύρια ευρώ. Και στην τελευταία θητή υπήρξε ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μιλάει για τις δαπάνες όσον αφορά το κλίμα και λέει ότι πρέπει να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 30% μέχρι το 2027 το αργότερο. Αυτά σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Ένα άλλο θέμα που εξετάζεται είναι ένα ταμείο δίκαιας μετάβασης που προτείνει ε, την καθαρή ενέργεια σε διάφορες περιοχές ε, που έχουν άνθρακα μέχρι τώρα και ζητάμε 4,8 δισεκατομμύρια για αυτό το ταμείο στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τους στόχους για τις εκπομπές είναι ότι από τη μία έχουμε το ETS, δηλαδή την διάθεση δικαιωμάτων ρήπανσης και από την άλλη μεριά έχουμε αυτούς που δεν συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό έχει ένα στόχο, μείον 21% για το 2020 και μείον 43% για το 2030. Και μέχρι το 2020 ο ρυθμός είναι ένα 0,74%, μείον 1,74% δηλαδή το χρόνο και θα φτάσει στο μείον 2,2%. Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει 45% των εκπομπών του θερμοκηπίου σε 11.000 εγκαταστάσεις και υπάρχει νομοθεσία για το τέταρτο στάδιο που εγκρίθηκε το 2018. Τώρα, πώς κατανέμονται τα δικαιώματα. Γίνεται ένας πληστηριασμός ή και ελεύθερα και στη δεύτερη περίπτωση αυτό ισχύει σε τομείς όπου υπάρχει ιδιαίτερος ανταγωνισμός στον κλάδο και πολλές πιθανότητες οι επιχειρήσεις, τα εργοστάσια να μεταγκατασταθούν αλλού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε και την εξή κατάσταση. Στο αρχικό στάδιο του προγράμματος αυτού διάθεσης δικαιωμάτων υπερβήκαμε τις εκπομπές. Υπήρξε ένα πλεόνασμα δηλαδή 2,1 δισεκατομμύρια τόνοι διοξιδίου του άνθρακα. Κάτι το οποίο οδήγησε βέβαια σε χαμηλότερες τιμές για τα δικαιώματα. Το πρώτο μέτρο μεταξύ 2014 και 2016 ήταν ένα backload, μια καθυστέρηση δηλαδή 300 εκατομμυρίων τόνων. Και τώρα στο νέο στάδιο υπάρχει ένα νέο μέσο που ονομάζεται το αποθεματικό σταθερότητας αγοράς ήδη από φέτος. Οπότε τα αποθέματα πηγαίνουν σε ένα αποθεματικό και τα δικαιώματα βγαίνουν από αυτό το αποθεματικό εφόσον οι δείκτες δείχνουν ότι πέφτουν τα δικαιώματα κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο. Και από το 2023 και μετά ο αριθμός των δικαιωμάτων σε, σε αυτή την αγορά θα περιοριστεί στα περσινά ποσά. Οι τιμές αυξάνονται πάντως στο πρόγραμμα ανταλλαγής δικαιωμάτων. Εδώ βλέπετε τα δικαιώματα και βλέπετε ποιες χρονιές είναι πιο ψηλά και πότε δεν είναι. Το κίτρινο κομμάτι είναι το συσσωρευμένο πλεόνασμα και η κόκκινη γραμμή δείχνει τις τιμές των δικαιωμάτων και ήδη βλέπετε εδώ το 2018 την αύξηση της τιμής μετά από το μέτρο αυτό εισαγωγής του αποθεματικού σταθερότητας της αγοράς από τον Ιούλιο που είμαστε στα 25 ευρώ περίπου τον Ιούλιο που μας πέρασε. Οπότε βλέπετε ότι συνεχίζεται η ενωδική πορεία. Τώρα, για το πρόγραμμα ανταλλαγής δικαιωμάτων ε, ρήπανθης. Εδώ πέρα ο στόχος ε, μείων 55% σε σχέση με το 1990 σημαίνει ότι η μείωση και μέσα στο πρόγραμμα ETS θα πρέπει να αυξηθεί. κάτω δηλαδή από το 2005 κατά 61 με 65% αντί για 43%. Και αυτό μπορεί να γίνει είτε με κύρωση δικαιωμάτων, είτε μέσω της ε, αγοράς, της ε, τοποθεματικού αυτού σταθερότητας αγοράς κλπ. Υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία που συμμετέχουν με εγκαταστάσεις στο ETS και οι εκπομπές αν δεν είναι στο ETS θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση με μεγάλο πλεόνασμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να κυρωθούν και άλλα δικαιώματα. Σε μερικές χώρες υπάρχουν τέτοιες ε, προτάσεις ήδη για να κυρωθούν τέτοια δικαιώματα. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται στις χώρες μέλη και όχι μόνο βέβαια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για κρατικές ενισχύσεις που εκπνέουν στα τέλη του 2020 και θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Είναι κάτι που υπάρχει στην ημερήσια διάταξη. Και στο τέταρτο στάδιο του ETS ε, προβλέφθηκε ένα ταμείο εξοχρινισμού. Αυτό είναι κάτι νέο ένα ταμείο το οποίο στηρίζει τις επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό των συστημάτων ενέργειας και την ε, ενεργειακή απόδοση. Θα υπάρξουν ετήσιες εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2024. Τώρα έχουμε και το άλλο κομμάτι που είναι οι εκπομπές εκτός συστήματος ανταλλαγής δικαιωμάτων ρήπανσης, εκτός ETS. Εδώ πέρα πρόκειται κυρίως για τις μεταφορές, για την κατοικία, γεωργία, απόβλητα. Εδώ η στόχη είναι μείον 10% για το 2020 και μείον 30% για το 2030, συγκρίνοντας με το 2005. Εδώ στο σκούρο μπλε ε, βλέπετε τις χώρες μέλη τι έχουν κάνει οι ενόψεις του 2020 και σε ανοιχτό μπλε τους στόχους για το 2030. Αυτό για να δείτε ότι οι στόχοι για το 2030 είναι πολύ πιο αυστηροί από ό,τι ήταν για το 2020 για πάρα πολλές χώρες. Όταν ε, βλέπετε τις σημερινές προβολές των χωρών μελών όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, υπάρχουν ε, λίγες χώρες. Αυτές που είναι σε πράσινο στο χάρτη αυτό, που ήδη εφαρμόζουν μέτρα για να πετύχουν τους στόχους του 2030 και σε πορτοκαλί είναι οι χώρες οι οποίες ακόμα βρίσκονται μακριά από την προβολή τους και τους στόχους εκτός συστήματος ETS. Εδώ είναι η αξιολόγηση. Έπρεπε έτσι κι οι χώρες να ε, παρουσιάσουν τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Και εδώ βλέπουμε ότι εκτός CTS, μεταφορές δηλαδή κατοικία και γεωργία, θα πέσουμε κάτω από το 2% σε σχέση με τους στόχους για το 2030. Και πολλές χώρες μέλη δεν παρουσίασαν τα σχέδια αυτά που δείχνουν τι γίνεται με το στόχο τους. Άλλε πάλι έχουν παρουσιάσει επιπλέον μέτρα. Υπάρχουν πάντω συστάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει οι χώρε μέλη να παρουσιάσουν αναθεωρημένα σχέδια μέχρι τα τέλη τη χρονιά αυτή. Κάτι το οποίο θα αξιολογηθεί και πάλι. Εδώ βλέπετε τους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι ένα πακέτο όπου έχουμε ένα στόχο του 20% ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 2020 και 32% ανανεώσιμες πηγές το 2030 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ Υπάρχει η οδηγία για τις ανώσιμες πηγές που προβλέπει η ρήτρα για την αναθεώρηση προς τα πάνω των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2023. Θα είναι δηλαδή στην ημερήσια διάταξη αυτής της θητείας. Και υπάρχει επίσης και η αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα των χωρών μελών όπου βλέπουμε ότι προς το παρόν υπάρχει μια διαφορά 1,1 με 1,6% για να πετύχουμε το στόχο του 32% από ανανεώσιμε πηγέ το 2030. Η επίτευξη του στόχου αυτού για το 2030 εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό από τη συνεισφορά των πιο φιλόδοξων χωρών μελών. Έχουμε επίσης στόχους και για την ενεργειακή απόδοση σε σχέση με την αρχική και την τελική σε σχέση με την αρχική είναι μείον 13%. 13%, 13% βελτίωση το 2020 και 26% το 2030. Και εδώ ε, στην αξιολόγηση των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα των χωρών μελών, εξακολουθεί να υπάρχει μια διαφορά όσον αφορά την επίτευξη του στόχου ενεργειακής επάρκεια ε, και απόδοση για το 2030, που είναι τη τάξης 2 με 6 ποσοστιαίες μονάδες. Μόνο λίγες χώρες μέλη έχουν ε, προσφέρει τη συνεισφορά του όσον αφορά την, ε, το στόχο αυτό τη ενεργειακή απόδοση. Εδώ βλέπετε τώρα τι συμβαίνει με την αεροπορία η διεθνή αεροπορία δεν συμμετέχει στον ευρωπαϊκό στόχο. Όσον αφορά δηλαδή τα αέρια του θερμοκηπίου. Και εδώ βλέπετε ότι στο εσωτερικό είναι σταθερή κάπως η κατάσταση, ενώ σε διεθνές επίπεδο υπάρχει μεγάλη αύξηση, γιατί η διεθνή αεροπορία 99% των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι από πτήσει οι οποίε ξεκινούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε έχει μεγάλο μερίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Εδώ πέρα έχουμε την ε, εξή κατάσταση. Οι χώρες γενικά έχουν συμφωνήσει σε διεθνέ επίπεδο έτσι ότι η Διεθνή Οργάνωση για την Οροπορία η ΚΑΟ, θα εκπονήσει μέσα και εργαλεία για τη μείωση των εκπομπών. Οι χώρες μέλη πρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να συνεργαστούν εξού και ο ΙΚΑΟ ανέπτυξε ένα πρόγραμμα αντιστάθμισης που το ονομάζει Κόρσια. Τις λεπτομέρειες δεν τις ε, έχουμε ακόμα, δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί πλήρως. Για παράδειγμα, ε, ποιες μονάδες θα συμμετέχουν ε, ή πώς θα υπάρξει συμμόρφωση με τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές ή με τη Συμφωνία των Παρισίων. Πάντω η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό Κόρσια ή κατά πόσο οι εκπομπέ από την αεροπορία θα συνεχίσουν να συμπεριλαμβάνονται ε, σε πρόγραμμα ETS. Είχαμε συμπεριλάβει στο ETS όλες τις εκπομπές από την αεροπορία, αλλά μετά υπήρξε μια άλλη πρόταση που έλεγε ότι το διεθνές κομμάτι δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί αλλά μόνο το κομμάτι των ETS μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πρέπει να δούμε τελικά τι θα αποφασιστεί και σε σχέση με τον ΙΚΑΟ. Έχουμε και άλλες συζητήσεις στην αεροπορία που λένε ότι η εμπορική αεροπορία ε, εξαιρείται από την ενεργειακή φορολόγηση. Κάποιες χώρες όμως έχουν επιβάλει φορολογία στην κυροσύνη και υπάρχουν και κατευθυντήριες γραμμές για τα αεροδρόμια και τις κρατικές ενισχύσεις. Η χρήση τώρα των ε, καυσίμων από εναλλακτικές πηγές ενέργειας στην αεροπορία αποτελεί μια πρόκληση. Και έχει να κάνει βέβαια και με την έρευνα που γίνεται, με την καινοτομία επίσης. Ερχόμαστε τώρα στην αυσιπλοεία. Οι διεθνεί νευσίπλοοι και εκπομπέ τη δεν συμπεριλαμβάνονται στου στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Απρίλιο του 2018 ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός συμφώνησε ένα αρχικό επίπεδο μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στόχοι είναι να μειωθούν ετησίως κατά 50% μέχρι το 2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 2008. Πρόκειται δηλαδή για έναν μακροπρόθεσμο στόχο. Βραχυπρόθεσμα μέτρα μένει ακόμα να αποφασιστούν υπό τον Διεθνή Νευτιλιακό Οργανισμό, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κανένα χρονοδιάγραμμα για τα μέσο ή μακροπρόθεσμα μέτρα. Όσον αφορά την οδηγία τώρα για το πρόγραμμα ανταλλαγής δικαιωμάτων ρήπανση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να αναθεωρείται τακτικά η δράση του Διεθνούς Νευτιλιακού Οργανισμού και ζητάει οι αδράσεις για να αντιμετωπιστούν οι εκπομπές στην ναυσιπλοεία και να το φροντίσει αυτό ίδιο ίδιος ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζουμε από το 2023, δεχομένω την προπαρασκευαστική δουλειά και τις διαβουλεύσεις. Υπάρχει βέβαια και το σύστημα συλλογής στοιχείων από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς τελικά θα λάβουμε υπόψη μας και τις εκπομπές της ναυτιλίας. Τώρα εδώ βλέπετε όπως είχαμε κάνει πριν για την αεροπορία και για την αυτιλία. Οι εκπομπές από την αυτιλία. Η πορτοκαλιά γραμμή είναι η βασική. Και μετά βλέπετε στη δικαιοκομένη μπλε ε, το σενάριο για υψηλή ζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν γι' αυτό να δούμε πώς θα έχουμε μέτρα μείωσης. Ένα άλλο τομέα τώρα που υπάρχει στην ημερήσια διάταξη είναι οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τα οχήματα. Υπάρχει η νέα νομοθεσία στη τελευταία θητεία, υιοθετήθηκε και ο κλάδος των μεταφορών έχει δείξει πολύ ψηλές εκπομπές και είναι υπεύθυνο για το 22% του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τα ΙΧ έχουν αυξήσει τις εκπομπές τους 120,4 γραμμάρια διοξίδιο του άνθρακα ένα χιλιόμετρο, ενώ ο στόχος για το 2020 είναι 95 γραμμάρια ανά διοξίδιο του άνθρακα. Είμαστε μακριά ακόμα δηλαδή. Βλέπουμε ότι οι πωλήσει υβριδικών οχημάτων ή ηλεκτρικών αυξάνεται πράγματι, αλλά το συνολικό μερίδιο της κατηγορίας αυτής ε, είναι χαμηλό, δηλαδή είναι ακόμα χαμηλά τα ηλεκτρικά ή τα υβριδικά σε πολλές χώρες Μόνο κάποιες εξαιρέσεις υπάρχουν όπως η Νορβηγία. Τώρα όσον αφορά την νομοθεσία, προβλέπεται αναθεώρηση του κανονισμού ε, που έχει να κάνει με τις επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, τον ε, ΙΧ για το 2023, όπως επίσης και για τα βαρέα οχήματα το 2022. Επίσης υπάρχει και οδηγία για την φόρτωση ε, βαρέων ε, φορτίων στα οχήματα. Για την περίπτωση αυτή πάλι θα υπάρξει, προβλέπεται μια αναθεώρηση για τη σχετική οδηγία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι χώρες ε, μέλη μπορούν βέβαια να βάζουν κάποια διόδια ανάλογα με την απόσταση αλλά ανάλογα και με το κόστος του φορτίου οι εκπομπές του διεξουδίου του άνθρακα πάντας και του αερίου του θερμοκηπίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέεται με το φορτίο. Τώρα, σε σχέση με τις προτάσεις της κυρίας Φοντερ Λάιεν και τις επιστολές, έγινε συζήτηση για ε, και έναν φόρο άνθρακα. Ένας τέτοιος φόρος δεν θα επέτρεπε τη μετεγκατάσταση εταιριών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο είναι γνωστό ως carbon leakage. Οπότε ένας τέτοιος φόρος θα μπορούσε να έχει να κάνει με τις αγωγές ή μείωση στις εξαγωγές. Πάντως έτσι να μπει κάποιο, κάποια τιμή, κάποιο δικαίωμα στις ε, χώρες εκείνες ή στις ε, επιχειρήσεις εκείνες που δρούν εκεί όπου δεν υπάρχει κάτι με το ETS. Πάντως προσπαθούμε με το ETS να αντιμετωπίσουμε αυτές τις περιπτώσεις. Η κλάδη, η οποία είναι εκτεθειμένη ε, στην δυνατότητα αυτή μεταγκατάστασης έχουν ε, ελεύθερα δικαιώματα. Δωρεάν. Άμα δείτε τις διάφορες ε, μελέτες, ε, πάντως δύσκολα αυτό συνάδει με τους κανόνες του ΠΟΕ. Ο φόρος τώρα στα σύνορα που λέγαμε σε σχέση με την μετεγκατάσταση και εδώ πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πραγματικότητα πως και τα δωρεάν δικαιώματα. Τελευταία μου διαφάνεια στις διάφορες συζητήσεις βέβαια μπαίνουν και τα ρηκτρά καύσωνα. Το 2009 οι επικεφαλείς του G20 συμφώνησαν να μειωθούν και να εξαφανιστούν τελικά τα ορυκτά, οι επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα μεσοπρόθεσμα. Και η πιο πρόσφατη έκθεση του Ενωρίου του 2019 δείχνει ότι οι ενισχύσει στα ορυκτά καύσωνα παραμένουν σταθερές ανάμεσα στο 2008 και το 2016 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν μειώθηκαν παρά των δεσμεύσεων σε διεθνές επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή είπε ότι θα αξιολογήσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη φορολόγηση της ενέργειας ώστε να ενισχυθεί αυτή η σταδιακή μείωση των ενισχύσεων. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε να αποκλειστούν ε, καύσιμα ε, με, τα χρήματα που βγαίνουν δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο του Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής για τα ορυκτά. Και εδώ ολοκληρώνω την παρουσίασή μου για τις μελλοντικέ προκλήσεις που είναι πολλές όπως βλέπετε. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητιέται και από το κοινό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. dokumentima. Mi u Hrvatskoj imamo problema s dokumentima.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 Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την πρώτη συγκεκριμένη ερώτηση για το κατεπόσο οι κανόνες παρακολούθησης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού επιτρέπουν συγκεκριμένα για τα εμπορευματοκιβώτια ή γενικά για το κάθε πλοίο. Αυτό πρέπει να το ελέγξω γιατί δεν έχω τις πληροφορίες για να σας τις δώσω τώρα. Όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε για, την, ε, για τον φόρο προσαρμογής άνθρακα. Όπως σας είπα, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τον ΠΟΕ, αλλά αυτό που πρέπει να δούμε είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής δικαιωμάτων ε, ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τα θέματα ανταγωνισμού. Ο, γι' αυτό και δίνει δωρεάν τα δικαιώματα σε εργοστάσια που υπόκεινται σε πολύ έντονο ανταγωνισμό. Ε, γι' αυτό δεν πληρώνουν, έχουν δωρεάν αυτά τα δικαιώματα. Και αυτό είναι ο τρόπος για να προστατεύσουμε αυτές τις βιομηχανίες, αυτούς τους κλάδους. Και εντάξει, δεν έχετε επιπλέον κόστο για να αγοράσετε τα δικαιώματα, γιατί ούτε και οι αντίστοιχοι κλάδοι άλλων χωρών ε, πρέπει να πληρώσουν για αυτά τα δικαιώματα. Οπότε έτσι μπαίνουν επίσης ώρες. Τώρα, επιπλέον μπορεί να υπάρχει ο φόρος προσαρμογής άνθρακα ή και δασμοί. Πρέπει να δει κανείς πώς συνδυάζονται όλα αυτά βέβαια και σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο θέμα να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγχρόνως και τα δύο εργαλεία. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ήθελα να πω ότι πρόκειται για εργαλείο πολιτικής, ότι ο πληστηριασμός είναι δηλαδή πολιτική. Απλώς είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα και μετά βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα ευθυγραμμιστούμε με τους κανόνες του ΠΟΕ. Τώρα συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε, ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αντιμετωπίσουμε τα θέματα διεθνούς ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, έχουμε σάγει κάτι το οποίο δεν το έβαλα στην ε, παρουσίασή μου, τον κανονισμό ΕΦΚΑ. Και οι εισαγωγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει αυτού έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως οι ευρωπαϊκοί κλάδοι για να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο μείωσης των εκπομπών και όλες οι εισαγωγές υποβάλλονται στον κανονισμό ΕΦΚΑ. Ευρωπαϊκές και μη. Οπότε ανάλογα με τον κλάδο είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε το θέμα του ανταγωνισμού. Πάντως το θέμα ε, προσαρμογής άνθρακα είναι μία ιδέα. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι. Έπειτα ρωτήσατε σε τι βαθμό οι ευρωπαϊκοί στόχοι ευθυγραμμίζονται με τον 1,5 βαθμό που είναι η έκθεση του IPCC και το σενάριο αύξησης θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό. Τα σενάρια της ε, IPCC δεν είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα για να ε, μας βοηθήσουν, γιατί έχουμε τις διάφορες χώρες, έχουμε και το παγκόσμιο επίπεδο, οπότε θα έπρεπε κανείς να καταφέρει από εκεί να μπει σε συγκεκριμένα σενάρια για κάθε μία χώρα. Πάντως, αν κοιτάξει κανείς γενικά τον προϋπολογισμό που στηρίζει και συνολικά και αναπεριφέρεια ε, το σενάριο αυτό του 1,5 βαθμού, Αυτό που έκανε το EPCC είναι ότι αύξησε τον προπολογισμό μέχρι το 2030. Ήταν αρκετά ε, γενναιόδωρο. Και μετά από το 2030 μέχρι το 2050 είναι πιο αυστηρό σε σχέση με τον 1,5 βαθμό. Με ρωτήσατε επίσης πώς να συμβιβάσουμε τις φιλοδοξίες για μείωση των εκπομπών με την καθοδική πορεία της οικονομίας. Αφενός έχουμε ανάγκη για πολλές επενδύσεις, από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε από το παρελθόν ότι η περίοδο κατά το παρελθόν όπου είχαμε μεγάλες περικοπές εκπομπών, η οικονομία ε, πήγαινε άσχημα. Οπότε αυτά τα δύο πρέπει να τα δούμε και συνδυασμένα. Άλλη ερώτηση. Με ρωτήσατε για τις επενδύσεις σε φυσικό αέριο και την μετάβαση που χρειάζεται και ρωτήσατε πετρέλαιο, άνθρακας, ε, ε, φυσικό αέριο. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο που χρειάζεται το φυσικό αέριο. Αλλά πάντως σε έναν κόσμο ουδέτερο αποτυπώματος άνθρακα το 2050 το φυσικό αέριο δεν θα έχει πια κανένα ρόλο να παίξει γιατί πρόκειται για ορυκτό καύσιμο. και άρα θα πρέπει να πάψουμε να έχουμε φυσικό αέριο. Άρα το ίδιο θα και με τις επενδύσεις για το φυσικό αέριο ότι θα πρέπει να εξαφανιστούν. Ρωτήσατε τώρα για τις τεχνολογικές προκλήσεις στο βιομηχανικό κλάδο. Αναφέρθηκε η αλλουργία. Υπάρχουν και άλλοι όπω όπως το τσιμέντο που εκπέμπουν ε, αέρια του θερμοκηπίου. Και είναι αλήθεια ότι στη βιομηχανία εξακολουθούμε να έχουμε ε, τεχνολογικές δυσκολίες, δηλαδή ότι δεν έχουμε όλες τις λύσεις που χρειαζόμαστε, συνεπώς χρειάζεται περισσότερη έρευνα στους κλάδους αυτούς της βιομηχανίας, ώστε να έχουν τελικά συστήματα παραγωγής χωρίς αέρια του θερμοκηπίου. Από την άλλη βέβαια έχουμε ήδη πρόοδο στην τεχνολογία, αρκετή. Χρειάζεται και άλλη, αλλά έχουμε αρκετή. Οπότε την καινοτομία ε, που έχουμε από την έρευνα πρέπει και να την εφαρμόσουμε στους βιομηχανικούς κλάδους. Να έχουμε μια πραγματικά καινοτόμο πολιτική. Πάντως είναι ένας τομέας όπου χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά και παραμένουν μπροστά μας πολλές προκλήσεις. Και έρχομαι τώρα στη δύσκολη πραγματικά ερώτηση. Δηλαδή, πώς να σταματήσουν οι κινητήρες καύσης και να υπάρχει αυτή η απαγόρευση στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ξέρω ότι περιμένετε την απάντησή μου. Αλλά μάλλον ξέρετε, γιατί και εσείς παρακολουθείτε από κοντά τι κάνουν οι χώρες μέλη με τους στόχους που θέτουν. Αυτό πάντως που βλέπουμε τώρα είναι ότι έχουμε κάποιους κατασκευαστές ε, αυτοκινήτων που δέχονται αυτούς τους στόχους και τους προωθούν. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα ότι δηλαδή η ίδια αυτοκινητοβιομηχανία ε, δεσμεύεται για τέτοιους στόχους. Αλλά κατά πρέπει να το συζητήσω περισσότερο με τους συναδέρφους μου που ασχολούνται με τις μεταφορές, γιατί εγώ δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις και έτσι ολοκληρώνουμε τον πρώτο γύρο της συζήτησης. Φυσικά απομένουν πολλά θέματα ακόμα, αλλά νομίζω ότι έχουμε μια επισκόπηση των ε, τομέων και θεμάτων ε, που θα συζητήσουμε αργότερα. Και βλέπω ότι ε, ήδη η συγγήτρια για την ναυτιλία σας έθεσε κάποιες ερωτήσεις, διότι γνωρίζει τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο Διεθνού Οργανισμού Ναυτιλίας και τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ευχαριστώ πολύ, Άνκε, που μας έθεσε στο πλαίσιο και περνάμε στην δεύτερη ομιλήτρια, Φρανσίσκα Βόλφ, επίσης από το Eco Institute. Να δούμε αν εσύ θα μπορέσει να περιοριστείς στα 15 λεπτά και στην επιστροφή σας μπορείτε να συγκρίνετε αποτελέσματα. Εσύ λοιπόν θα μας παρουσιάσεις ε, την κατάσταση και τις προκλήσεις ε, στην πολιτική περιβάλλοντος. Σε ευχαριστώ Μπας για την εισαγωγή σου. Εγώ θα ε, καλύψω πολλά θέματα, τα περιβαλλοντικά που δεν έχουν να κάνουν με το κλίμα, ε, το οποίο σημαίνει ότι ε, μπορεί να δυσκολευτώ να ε, παραμείνω εντός του 15 λεπτού, αλλά κάποια θέματα έχω επιλέξει να αναφέρω. Πολλά άλλα θέματα έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της περασμένης θητείας. Η ε, δομή της ε, μελέτης ε, μου, της παρουσίασής μου είναι παρόμοια με της συναδέρφου. Θα ξεκινήσω από κάποια γενικά θέματα και θα προχωρήσω κατόπιν σε κάποια που έχουν συμπεριληφθεί στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις τελευταίες εβδομάδες. Κατόπιν θα προχωρήσω σε κάποια θέματα όπου διαπιστώθηκαν κενά στην εφαρμογή. Θα καλύψω θέματα που προβλέπεται να επανεξεταστούν ε, και λόγω της νομοθετικής διαδικασίας για τα θέματα που θα καλύψω. Θα σας δώσω πρώτα κάποιες σύντομες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση, ε, σε τι στάδιο βρίσκεται η συζήτηση, αλλά κατόπιν ε, και θέματα που έχουν εντοπιστεί και από το Κοινοβούλιο και από άλλα θεσμικά όργανα για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε τα θέματα αυτά. Όσον αφορά τα γενικά θέματα, υπάρχουν διάφορες ε, προκλήσεις και προβληματικές τάσεις, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, στην επόμενη νομοθετική περίοδο. Έχουμε τα νητρικά, τα απόβλητα, την ε, ρήπανση, ε, σε τρεις βασικές ομάδες όμως μπορούμε να ε, τα μοιράσουμε αυτά, την κατανάλωση πόρων, ε, την ε, ποιότητα του περιβάλλοντος και τη βιοπικιλότητα. Η βασική στόχη για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι λείπει μια γενική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης με αναλυτικά χρονοδιαγράμματα, στόχους, θεσμικές δομές κλπ. Το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να προσανατολίζεται περισσότερο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και πέρα από τα οικονομικά θέματα πρέπει οι ε, περιβαλλοντικές ανησυχίες να ληφθούν υπόψη σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περιβαλλοντικές πολιτικές ε, χρειάζονται επίσης καλύτερη χρηματοδοτική βάση. έχει παρατηρηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον όσον αφορά την προστασία του ε, φυσικού κεφαλαίου, τη βιοπικιλότητα. Ε, επίσης ε, δεν είμαστε πολύ αποτελεσματικοί ως προς τους πόρους και ιδιαίτερα η ποιότητα των υδάτων είναι σημαντικό θέμα όσον αφορά την ενσωμάτωση των ε, περιβαλλοντικών ε, πτυχών ε, σε διάφορες πολιτικές, την κοινή γεωργική πολιτική, την κοινή πολιτική αλληλείας, είναι θέματα που μας απασχολούν, όπως επίσης στα διαρθρωτικά ταμεία και στην πολιτική συνοχής. Τα καλά νέα όπως γνωρίζετε, είναι ότι η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φοντερ Λάιεν ε, προτείνει ε, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των πρώτων 100 ημερών ε, της θητείας της. Ε, που περιλαμβάνει πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα, όπως είναι η δέσμευση για κλιματική ουδετερότητα, ένα νέο ταμείο δίκαιης μετάβασης ε, που θα στηρίξει βιομηχανίες ε, που επηρεάζονται αρνητικά από τις νέες πολιτικές, μια στρατηγική βιοπικιλότητας για το 2030, μια πολιτική μηδενικής ρήπανσης και μια, ένα νέο σχέδιο για κυκλική οικονομία που θα συμπεριλαμβάνουν τα μικροπλαστικά και μια νέα στρατηγική από ε, την ε, γεωργική εκμετάλλευση στο τραπέζι του καταναλωτή. Όσον αφορά λοιπόν το πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί η σχέση ανάμεσα στο Green Deal, αυτήν την πράσινη συμφωνία της Φοντερ Λάιεν, και το επόμενο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, που ε, θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων ήδη τώρα από το φθινόπωρο. Όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη, μετά από την ε, υιοθέτηση των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης το 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα, ε, μια γενική δέσμη μέτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνει ένα μακρόπνο όραμα και παρουσιάστηκαν τρία ε, σενάρια για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σχετικό ψήφισμα ε, επέλεξε, προτίμησε το πιο φιλόδοξο από τα τρία αυτά σενάρια και προτείνει η υιοθέτηση μια γενική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για εφαρμογή των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη με αναλυτικά χρονοδιαγράμματα ε, μέχρι το 2030. Και επίση συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένε προτάσει για τι θεσμικέ δομέ και ένα πλαίσιο για να ε, ε, διασφαλιστεί η συμπέληψη των πολιτικών αυτών στην νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, ε, το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο θέλουν ε, ε, τα, οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη να συμπεριλαμβάνονται στι πολιετή προτεραιότητε των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι τομεί όπου το Κοινοβούλιο διαπίστωσε ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω δουλειά και που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι οι παγκόσμιε αλυσίδε αξία, οι κάτι που σχετίζεται με επιχειρήσεις ε, αλλά και με ανθρώπινα δικαιώματα, ε, την βιωσιμότητα σε εμπορικές συμφωνίες, σε ένα πλαίσιο ε, βιώσιμων επενδύσεων, βιωσιμότητα στα εισαγόμενα προϊόντα όπως είναι το φινικέλαιο, τα βιοκάψιμα κλπ. και ε, βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και κατανάλωση. Και η τελευταία μου διαφάνεια σε αυτό το κεφάλαιο είναι ότι όλοι γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα νέο πρόγραμμα LIFE ύψους 5,45 ε, δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την ε, τελευταία θητεία πρότεινε να αυξηθεί στα 7,27 ε, δισεκατομμύρια η χρηματοδότηση και ζήτησε επίσης συμπερίληψη των περιβαλλοντικών πολιτικών στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, σε όλους τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού και προτείνει επίσης υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση της λειτουργίας του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Επίσης ε, προτείνει τη δημιουργία ενός ε, Ταμείου Δίκαιης Ενεργειακής Μετάβασης, σε κάτι που ήδη έκανε η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν και να αποκλειστεί η παραγωγή ορυκτών καυσίμων ε, και η μηχανές εσωτερικής ανάφλεξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. Κάποια θέματα αναφέρθηκαν συγκεκριμένα από την νέα πρόεδρο στο θεματολόγιο της για την Ευρώπη και ε, στις επιστολές ε, ε, της αποστολής της στους επιτρόπους Τίμερμανς και Βιτσούτης. Και Ένα από αυτά σχετίζεται με την χρήση γης και το εθνικό κεφάλαιο. Όλοι γνωρίζετε τον έλεγχο καταλληλότητας της ε, οδηγίες για τα ύδατα και για τους ε, βιότοπους και οι δύο αυτές οδηγίες παραμένουν σημαντικές. Ε, θα πρέπει όμως να ενισχυθούν. Τα δίκτυα Natura 2000 είναι ακόμη ατελή στα περισσότερα κράτη-μέλη και υπάρχει έκθεση για την αναχέτηση της της απώλειας ε, ε, ε, διοπικιλότητας από την Ευρώπη. Επιλογές για να αντιμετωπιστούν περαιτέρω προκλήσεις. Η ενσωμάτωση πτυχών διοπικιλότητας σε άλλες πολιτικές, όπως είναι η κοινή γεωργική πολιτική, αλλά και την κοινή πολιτική αλίας, καθώς και άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε επίση ε, να ενισχυθεί η χρηματοδότηση για την ε, βιοπικιλότητα στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, να ε, έχουμε αναβίωση τη πολιτική για την ποιότητα του εδάφου, κάτι που εγκαταλείφθηκε το 2014 νομίζω, μπορεί όμω να ξαναξεκινήσει τώρα με την δημοσίευση της έκθεσης της IPCC που τονίζει την ποιότητα της τη σημασία της ποιότητας του εδάφους για το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την ε, διατροφική ασφάλεια. Επίσης, η στρατηγική βιοπικιλότητα θα πρέπει να στηρίζεται από στόχου ε, και ε, χρηματοδότηση, όπως ζήτησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και προτάθηκε επίσης να βελτιωθεί η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την ξυλία, καθώς και να αυξηθεί η συμμετοχή στην Σύμβαση για την βιοπικιλότητα που αυτή τη στιγμή ε, θεσπίζει το πλαίσιο που θα διαρκέσει μέχρι το 2030 όσον αφορά την ε, αποδοτικότητα των πόρων, την κυκλική οικονομία και την ε, διαχείριση των αποβλήτων. Είχαμε το 2015 ένα σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που συνοδεύτηκε από διάφορες νομοθετικές προτάσεις. Έχουμε την ε, οδηγία οικολογικού σχεδιασμού που ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη οποία η αναθεώρηση ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη το 2015. Η κυρία Φοντερ Λάιεν ε, έχει ανακοινώσει τώρα ένα νέο σχέδιο δράση για την κυκλική οικονομία και άλλο σημαντικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά στην κυκλική οικονομία ε, πλέον έχει τεθεί σε ισχύ. Μελλοντικέ προκλήσει και πώς μπορούμε να σε αντιμετωπίσουμε. Να βελτιώσουμε την εφαρμογή της στρατηγικής για την κυκλική οικονομία, κάτι που αποτελούσε μέρος ε, της ε, έκθεσης ε, εφαρμογής της Κομισιόν. Να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό πέρα από τα προϊόντα που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας και να έχουμε κριτήρια για την αποδοτικότητα των πόρων. Επίσης, να διασφαλίσουμε, να εισάγουμε νέες απαιτήσει ώστε να έχουμε προϊόντα ε, μακράς ε, διαρκείας, ε, επίσης να χρησιμοποιούμε τα δευτερεύουσες πρώτες ύλες, να έχουμε ελάχιστα πρότυπα για την ανακύκλωση συγκεκριμένων πλαστικών, να απαγορεύσουμε τα μικροπλαστικά και τα καλλιτικά, και τα καλλιτικά που τα περιέχουν μέχρι το 2020, ε, επίσης, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των ανακυκλωμένων πλαστικών ε, και να έχουμε νομικά δεσμευτικούς ε, ορισμούς και στόχους για τα απόβλητα, καθώς και να αναθεωρήσουμε την οδηγία για τα, για τα παλαιά οχήματα. Η έκθεση του 2015 εντόπισε κάποια κενά στην... του 2019, συγγνώμη, εντόπισε διάφορα κενά στην εφαρμογή. Όσον αφορά τα τοξικά και τα φυτοφάρμακα, η νομοθεσία REACH λειτουργεί πλήρως, είναι πλήρως σε ισχύ από το 2018 και μετά. Η πρώτη έκθεση ε, εφαρμογής ε, αναμένεται το 2021. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει ε, στρατηγική για να προωθήσουμε κύκλο, ανακύκλωση για τα μη τοξικά υλικά. Ε, επίσης υπάρχει κενό όσον αφορά τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες ε, στα καλλιντικά, τα παιχνίδια και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Προτάσεις για να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις είναι να συμπεριληφθούν όλες οι οι ουσίες υψηλής ανησυχίας ε, στον ε, κατάλογο υποψηφίων ε, ουσιών για το REACH. Επίσης, να βελτιώσουμε τη συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH και να ενισχύσουμε τους συνοριακούς ελέγχους για να εμποδίσουμε την εισαγωγή απαγορευμένων ουσιών στην εσωτερική αγορά. Συγκεκριμένα όσον αφορά τα φυτοφάρμακα, προτάθηκε να βελτιωθεί το σύστημα αδειοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης να βελτιωθούν τα πρότυπα για την παρακολούθηση της χρήσης τους. Να εισαχθούν στόχοι για μείωση της χρήσης τους, να αυξηθεί η διαφάνεια της ε, διαδικασίας αδειοδότησης, ε, για παράδειγμα, δημοσιεύοντας τις μελέτες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Ζητήθηκε το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να κινητοποιήσει την ε, καινοτομία στα φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου και να παρέχονται δεδομένα για ε, την τοξικότητα των ε, ουσιών. Όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, ε, ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση μέχρι το 2020 για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες στα καλλιντικά, τα παιχνίδια και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και να επιταχυνθεί η διαδικασία δοκιμής και Έγκριση ε, των ε, ουσιών αυτών. Όσον αφορά τα μικροπλαστικά, ζητήθηκε απαγόρευσή τους σε κάποια προϊόντα και ζητήθηκε και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών ε, να εξετάσει το ενδεχόμενο απαγόρευση για μικροπλαστικά που προστίθενται σε άλλα προϊόντα. Είχαμε μια αντίδραση στις αρχές του 2019 όπου ζητήθηκε απαγόρευση για ε, επαγγελματική χρήση ε, για τα καλλιντικά για... και διάφορα άλλα προϊόντα. Όσον αφορά την ηχορύπανση, υπάρχει κάποια ε, νομοθεσία. Έχουμε όμως ε, υψηλά επίπεδα θορύβου στα αεροδρόμια από ε, μη υπερηχητικά στρατιωτικά αεροσκάφη, από αυτοκίνητα. Δεν έχει προταθεί καμία νομοθετική δράση παρά επανειλημμένα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει νομοθεσία για να μειωθούν τα επίπεδα θορύβου και να Επίσης έχουμε έλλειψη των σχεδίων δράσης ε, των κρατών μελών για τη διαχείριση του θορύβου και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό. Όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον, έχουμε ανεπαρκή δεδομένα ε, κάτι που δεν μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε την κατάσταση κάποιων θαλάσσιων περιοχών. Στο μέλλον, η αναθεώρηση της κοινή ε, πολιτικής αλληλείας αναμένεται το 2022. Και η νέα πρόεδρος Φοντερ Λάιεν αναφέρθηκε όχι μόνο σε μείωση της αλληλείας, αλλά και σε προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Ε, σε παγκόσμιο επίπεδο έχει συμφωνηθεί να απαγορευτεί η υπεραλίευση και να καταπολεμηθεί η ε, παράνομη αλληλεία. Ε, το 2020 θα πραγματοποιηθεί στην Λισαβόνα διάσκεψη των, ωκεανών, διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς. Επίσης κάποια θέματα τα οποία ούτως ή άλλως πρέπει να αναθεωρηθούν σύμφωνα με την κανονική νομοθετική διαδικασία είναι η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Έχουμε τη σχετική οδηγία η οποία αυτή τη στιγμή αναθεωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο έλεγχο καταλληλότητα ε, τη νομοθεσία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλο του 2019 και θα ακολουθήσει λογικά ε, σχετική νομοθετική πρόταση. το προηγούμενο κοινοβούλιο πρότεινε να ε, προωθηθεί η παραγωγή καθαρής ενέργειας ε, και να έχουμε τηλεθέρμανση για βελτίωση της ποιότητας του αέρα και επίσης να αντιμετωπιστούν τα κενά στην εφαρμογή ε, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Όσον αφορά τα ύδατα, Υπάρχει μια πρόταση για μια αναθεωρημένη οδηγία για το πόσιμο νερό. Ο τριμερής διάλογος αναμένεται να πραγματοποιηθεί τώρα το φθινόπωρο και το ίδιο ισχύει για μια πρόταση για κανονισμό για ελάχιστα, ε, ελάχιστες απαιτήσει για την επαναχρησιμοποίηση ε, υγρών αποβλήτων. Ε, και επίσης έχουμε πρόταση για αναθεωρημένη ε, ε, οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα που αναμένεται το 2021 όσον αφορά τις προκλήσεις αυτές. Έχει προταθεί ε, η οδηγία για το πόσιμο νερό να καλύπτει και άλλες ουσίες που σχετίζονται με την ασφάλεια του πόσιμου νερού. Μέγιστα όρια για κάποιους ε, ρήπους ε, και μικρόβια και θα πρέπει να έχουμε στη μέση για τις περισσότερες ρηπογόνες ουσίες, ενώ θα πρέπει να αυξηθεί η διαφάνεια για τους καταναλωτές. Επίσης, ε, οι στόχοι που σχετίζονται με το νερό θα πρέπει να ενσωματωθούν σε άλλες ε, τομεακές πολιτικές, όπως είναι η κοινή γεωργική πολιτική. Η επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων ε, θα πρέπει να ενισχυθεί. Και εκτός του αγροτικού πλαισίου. Ενώ η οδηγία για ε, την ε, ε, επεξεργασία των αστικών υδάτων θα πρέπει επίσης να ανεθεωρηθεί. Αυτά έχουν προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από άλλους ενδιαφερόμενους. Όσον αφορά την βιώσιμη χρηματοδότηση, θα γνωρίζετε ότι είχαμε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου που εκπώνησε έκθεση το 2018 και τα συμπεράσματα έχουν μετατραπεί σε νομοθετικές προτάσεις. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση και έχει υποβάλει μια σειρά από προτάσεις ε, σχετικά με το πώς αυτές οι νομοθετικές προτάσεις ε, του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να ενισχυθούν. Για παράδειγμα, το σύστημα ταξινόμησης για τις ε, βιώσιμες ε, οικονομικές δραστηριότητες ε, θα πρέπει να διευρυνθεί και το πλαίσιο θα πρέπει να καθορίζει και το επίπεδο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Συγγνώμη, λέει η ομιλήτρια, μπερδεύτηκα. να καθοριστούν κριτήρια για το πότε και πώς ε, οι οικονομικές δραστηριότητες έχουν αρνητικές συνέπειες στη βιωσιμότητα. Και επίσης να έχουμε εναρμονισμένα συγκρίσιμα και ενιαία κριτήρια και δείκτες λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της αλυσίδας αξίας ε, και να ε, εξετάζουμε και τον συνολικό κύκλο ζωής των προϊόντων. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από προτάσεις για την βιώσιμη οικονομία και τέλος για την κοινή γεωργική πολιτική. Όπως μάλλον όλοι γνωρίζετε, τρεις νομοθετικές προτάσεις ε, ε, υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018, το στρατηγικό σχέδιο της κοινή γεωργικής πολιτικής, τον οριζόντιο κανονισμό και τον τροποποιητικό κανονισμό. Η Επιτροπή Άγκρη ε, δημοσίασε έκθεση για το στρατηγικό σχέδιο ε, της κοινή γεωργικής πολιτικής με 109 τροπολογίες, οι οποίες όμως δεν έχουν ψηφιστεί ακόμα. Κάποιες από τις βασικές επικρίσεις ή προτάσεις ε, ήταν ότι οι άμεσες πληρωμές ε, θα πρέπει να ε, υποβάλλονται ε, ακόμη περισσότερο σε ρεσιμότητα και περιβαλλοντικούς στόχους στον πυλώνα 1. Στον πυλώνα 2 θα πρέπει τα διεθνή ποσά για εθελοντικά προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού. Επίσης, το ελεγκτικό συνέδριο Ε, Είπαν ότι ε, κάποιες προτάσεις δεν ήταν κατάλληλες για να πετύχουμε τους ε, κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον. Και άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν να συμπληρώσουμε την κοινή γεωργική πολιτική με μια κοινή πολιτική τροφίμων. Πολλά είπα. Νομίζω ότι ξεπέρασα και το χρόνο ομιλίας μου. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Thank you very much and, and only slightly missed the, the... Ναι, παραλίγο το τέταρτο, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Ορισμένες φορές ξεχνάμε ότι εκτός από το κλίμα υπάρχει και ένα τεράστιο περιβαλλοντικό θεματολόγιο. Μας δώσετε μια σαφέστατη εικόνα σε 20 λεπτά, πράγμα καθόλου εύκολο. Ερωτήσεις παρακαλώ. Η κυρία Πάουλης από ό,τι βλέπω από τους Πρασίνους θέλει να κάνει ερώτηση. Τρεις ερωτήσεις είναι, όχι μία. Ίσως ε, δεν ε, το είπατε, νομίζω ότι υπάρχει ένα σημαντικό θέμα που αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα στο νερό. Ε, από απόβλητα, επιφανειακά ύδατα, πόσιμο νερό κλπ. Και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον έχετε κάποια πρόταση να μας κάνετε για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο. Μετά, για την ανακύκλωση των πλαστικών. Το πρόβλημα που έχουμε, ή τουλάχιστον αυτό λένε οι παράγοντες της αγοράς, ότι λόγω της παρουσίας τοξικών ουσιών στα πλαστικά πολλοί προμηθευτέ δεν θέλουν να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο πλαστικό, γιατί αν θέλουν, ε, λένε ότι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πλαστικό για τη συσκευασία τροφίμων, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ ανακυκλωμένο ε, πλαστικό, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να περιέχουν. Και επίση υπάρχουν ε, ε, πλαστικά πολλαπλών επιπέδων, τα οποία δεν μπορούν να τύχουν ε, σωστού εις ανακύκλωση. Υπάρχει μια, κάποια άλλη προσέγγιση, για παράδειγμα, από τους μεγάλους παραγωγούς, ε, οι οποίοι εξετάζουν έναν τρόπο ανακύκλωσης πλαστικών σε πρώτες ύλες και ε, ε, να πάρουν κάτι αντίστοιχο ε, με το ε, ναύτα και να καταστρέφονται όλες οι ταξικές ουσίες. Γιατί μέχρι τώρα τα πλαστικά πολλών επιπέδων μπορούν απλώς ε, να περάσουν από διαδικασία καύσης. Κάτι το οποίο φυσικά δεν βοηθάει καθόλου και την κλιματική αλλαγή. Και μια τελευταία ερώτηση. Από ό,τι έμαθα πολλές από τις παρατάσεις που δίνονται για τα ζυζανιοκτώνα είναι γιατί τα κράτη-μέλη αργούν στην αξιολόγηση Αυτό που γίνεται είναι ότι η εταιρεία παραγωγή του φυτοφαρμάκου κάνει αίτηση, το κράτο μέλο πρέπει να κάνει αξιολόγηση και αν καθυστερήσει η αξιολόγηση δίνεται αυτόματα παράταση. Θα ήθελα να ξέρω πώ μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτό, διότι ε, είναι ζωτική σημασία να σταματήσουν αυτές οι πάρα πολύ επιζήμιες ουσίες, ε, να μην ε, ε, κυκλοφορούν στην αγορά ε, συνεχώς. Ευχαριστώ. Κυρία Βάης. Ναι φαντάζομαι εξακολουθεί να ισχύει το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχουν στοιχεία στις ερωτήσεις μου. Ναι, προσπαθήστε να το κάνετε αυτό. Ίσως ε, θα μπορούσε να είναι και νέο πρότυπο για πολλούς άλλους. Όσον αφορά την ε, οδηγία για τα οικολογικά, τι περίπτωση υπάρχει στο μέλλον να συμπεριληφθούν και πληροφορίες για το αποτύπωμα του άνθρακα προς τους καταναλωτές, αλλά και να θεωρηθεί και νέος τρόπος να ε, λαμβάνεται υπόψη από τους παραγωγούς για τον τρόπο με τον οποίο ε, παράγουν τις τεχνολογίες τους, ώστε να υπάρχει χαμηλότερο αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα. Όταν θα γίνει η επόμενη αναθεώρηση της οδηγίας ε, αυτής, ίσως θα μπορούσε να συμπεριληφθεί κάτι τέτοιο στη διαδικασία ή θεωρείτε ότι είναι καλύτερο να υπάρξει και μία ακόμα επισήμανση επί του προϊόντος ε, που θα έχει ένα σαφές μήνυμα και σαφή γλώσσα για το αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα για οποιοδήποτε προϊόν. Ευχαριστώ. Mr. Wallace. Thank you very much. Ο κύριος Wallace, ευχαριστώ πολύ. Αναφερθήκατε στην ε, νέα πράσινη συμφωνία της Βάντερ Λάιεν για την ε, ε, διαφάνεια για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, στην Ιρλανδία έγινε ολόκληρη συζήτηση γιατί οι μικρές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα, ζητάνε να υπάρχει καθαρότερη παραγωγή ε, κρέατος, πιέζονται από τις μεγάλες παραγωγές, οι μεγάλοι παραγωγοί κυριαρχούν στην αγορά και υπάρχει τεράστια έλλειψη διαφάνειας αυτή τη στιγμή όμως ε, για πάρα πολλά ε, στοιχεία ε, για το πώς φτάνει κάτι από το χωράφι στο τραπέζι μας, ακόμα και για την τιμολόγηση. Και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον σε αυτή τη νέα συμφωνία θα έχουμε και διαφάνεια για το τελικό ε, τρόφιμο τελικά. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, ε, αυτή τη στιγμή γίνεται εισαγωγή του 6,5 εκατομμύρια πέρσι, κυρίως από τη Λατινική Αμερική, ε, και πολλά από αυτά έχουν γενετικώ τροποποιημένους οργανισμούς, αλλά αν αγοράσεις ε, ε, μία συσκευασία βούτυρο στην Ιρλανδία, δεν λέει ότι το προϊόν αυτό μπορεί να περιλαμβάνει γενετικώ τροποποιημένους οργανισμούς, ενώ θα έπρεπε να το λέει. Και δεν ξέρω αν η κυρία Βέντερ Λάιεν αναφέρεται στο θέμα αυτό στην πρωτοβουλία. Σημαίνει επίσης ότι θα υπάρχει υποχρέωση διαφάνειας για το τι ακριβώς περιλαμβάνεται σε αυτά που τρώμε. Ε, διότι αυτή τη στιγμή η επισήμανση είναι ανεπαρκής ε, για να αντιμετωπίσουμε ε, προϊόντα χαμηλής ποιότητας και κρέατα τα οποία εισάγονται από τη Βραζιλία και επηρεάζουν την ποιότητα των τροφίμων μας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απλώ να τονίσω ότι εδώ έχουμε κόσμο από το Ινστιτούτο Όγκο, Επομένω δεν μπορούν να προβλέψουν και να μας πούνε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν το αναδιατυπώσετε βέβαια λίγο θα μπορούσατε να ρωτήσετε τι πιστεύετε ότι θα σημαίνει αυτή η διαφάνεια στην αλυσίδα τροφίμων. Έτσι ε, νομίζω ότι μπορεί να απαντήσουν και οι εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Όγκο. Ευχαριστώ. Πολλά έχουν υποθεί μέχρι τώρα και πολλά έχουν γίνει. Βέβαια υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις, αλλά κάτι αφήνουμε απ' έξω. Έχουμε δύο κρίσεις σήμερα. Η κλιματική αλλαγή είναι μία που συνεχίζεται, αλλά στη σκία αυτής της κρίσης υπάρχει και η κρίση της απώλειας βιοπικιλότητας παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι χάνουμε μορφές ζωής και χάνονται επειδή δεν έχουν τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να συνεχίσουν να ζουν. Χάνουμε λοιπόν ζωή όταν δεν μπορεί να προσαρμοστεί και αυτό αποτελεί μια οξία απειλή σε βάρος όλων μας. Αναρωτιέμαι τώρα Επίσης, για αυτή τη μαγική λέξη βιωσιμότητα, μιλάμε για βιώσιμη γεωργία, για βιώσιμη βιομηχανία, ναι, αλλά χάνουμε μορφές ζωής. Άρα, κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε για να διαχειριστούμε ε, την ε, ζωή αυτή. Αναρωτιέμαι, υπάρχουν εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να κάνουμε μια πιο σε βάθος αξιολόγηση της λεγόμενης βιωσιμότητας. Πολύ θα ήθελα να είχαμε ένα τέτοιο εργαλείο. Ευχαριστούμε. Τελευταία ερώτηση και μετά θα κάνω κι εγώ μία έτσι για να την κάνω. Η κυρία Βόλαντεν, συγγνώμη, πώς προφέρετε το όνομά σας. Βόλτεν. Ε, είναι γερμανικό, αν και εγώ είμαι Βρετανίδα. Ε, μερικές φορές είναι πιο εύκολο από ό,τι νομίζει κανείς. Παρακαλώ. Είμαι νέα Ευρωβουλευτής εδώ, νέα και στην Επιτροπή αυτή, δεν έχω πολύ καιρό που ασχολούμαι με αυτά. Θέλω όμως να ρωτήσω το εξής. Έχουμε ήδη, ακούσαμε την κρέτα του στη Νέα Υόρκη, ε, ακούμε και από χτες για το λιώσιμο των πάγων της Ανταρκτικής κτλ. Οπότε εγώ θέλω να μάθω περισσότερα ε, θα έπρεπε όντως να νιώθουμε απελπισμένοι με την ε, κατάσταση αυτή. Και επειδή είμαι σε μη κυβερνητική οργάνωση, θα ήθελα να ξέρω, πιστεύετε ότι κάνουμε αρκετά, πιστεύετε ότι παίρνουμε αρκετά στα σοβαρά τα προβλήματα αυτά. Σε κάθε επίπεδο θα πρέπει να έχουμε ριζοσπαστικές πολιτικές και αλλαγές για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ρε, καθόμαστε και σκεφτόμαστε τα πάντα, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε τα σοβαρά προβλήματα. Θα έπρεπε σε κάθε τομέα, γεωργία, εμπόριο, οικονομία, παντού. Θα ήθελα τη σκέψη σας. Ξέρω ότι δεν μιλάτε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα ήθελα να ξέρω τη γνώμη σας. Ε, πάντα όντω μπορούν να προσπαθήσουν κάτι να πούνε. Λοιπόν, η δικιά μου ερώτηση, λέει ο πρόεδρο, όταν μιλάμε για την κυκλική οικονομία. Είπατε και στην παρουσίασή σας ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, δηλαδή και το θέμα των πρώτων υλών και πώς ε, τις ε, πρώτες ύλες τις ε, επανακτούμε από χρησιμοποιημένα υλικά. Τι προτάσεις έχετε στο μυαλό σας εσείς για να βελτιωθεί αυτή η ανάκτηση των πρώτων υλών. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Δεν ξέρω, κανείς άλλος, τελευταία ευκαιρία για ερώτηση. Ωραία, η απάντηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, αυτό είναι το σημείο που πρέπει να ομολογήσω ότι ήμουνα ε, μία από τους τελευταίους που ασχολήθηκε με αυτή την έκθεση, που σημαίνει ότι για πολλά θέματα δεν είμαι ειδική και ειλικρινά είχα ε, ότι θα με ρωτήσετε για χημικά. Και να, που ο φιάλτης μου επαληθεύεται. Λοιπόν, πολλοί συναδελφοί μου έχουν ασχοληθεί με την χημική τη πολιτική απέναντι στα χημικά. Δεν είμαι ένας από αυτούς. Οπότε τι ερωτήσει σα θα πρέπει να τις περάσω στους συναδέρφους και αν μου αφήσετε το email σας θα τους ζητήσω να σας απαντήσουν ε, με email. Τώρα υπήρξε μία πτυχή... Η τρίτη από την πρώτη δέσμη ερωτήσεων είχε να κάνει με τα φυτοφάρμακα. Ότι παραμένουν στην αγορά ενώ η αξιολόγηση ε, δεν έρχεται έγκαιρα. Χωρίς αξιολόγηση δηλαδή. Και ρωτάτε τι πρέπει να κάνουμε. Ε, πρέπει να έχουμε περισσότερο προσωπικό τελικά στις αρχές που προβαίνουν στην έγκριση. Αυτή είναι μια ανησυχία που υπάρχει και σε πολλές χώρες μέλη, ότι δηλαδή οι διαδικασίε έγκριση είναι χρονοβόρες εάν γίνονται καλά και δεν έχουν αρκετό προσωπικό. Χρειάζεται χρηματοδότηση. Και αυτή ήταν μια έκκληση που έκαναν πολλοί ευρωβουλευτές στην προηγούμενη θητεία. Περισσότερα κονδύλια. Κονδύλια και για τις αρχές που έχουν ως εντολή να προβαίνουν στις αξιολογήσεις αυτές. Τώρα, το αποτύπωμα άνθρακα και πώς ε, συμπεριλαμβάνεται στην οδηγία για τον ε, οικολογικό σχεδιασμό. Αν ε, αυτό πρέπει να γίνει, αν χρειάζεται κάποιο νέο σήμα. Ούτε αυτό είναι δικός μου τομέας. Μπορεί να σας απαντήσω Λάθο. Πάντως η αίσθηση που έχω είναι ότι η ενέργεια και ο ανθρακάς είναι θέματα τα οποία καλύπτονται πολύ καλά από την οδηγία για τον οικολογιακό σχεδιασμό. Ε, και πάλι το θέμα έχει να κάνει με την ε, ενεργειακή απόδοση περισσότερο. Επίσης, ο οικολογικός σχεδιασμός ακριβώς έχει να κάνει με την απόδοση, δεν έχει να κάνει με απόλυτες τιμές ε, κατανάλωσης. Το θέμα δεν είναι ότι παράγουμε να γίνει όσο γίνεται πιο αποδοτικό, αλλά να έχουμε ε, ένα προϊόν το οποίο καταναλώνει πολύ χαμηλές τιμές. Απόλυτα, σε απόλυτες τιμές. Και εδώ, όπω είπατε και εσείς, δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως, πιστεύω ότι είναι must τέτοιες πληροφορίες για τα τελικά προϊόντα, κατά πόσο περιλαμβάνουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή βασίζονται σε αυτούς, ότι θα πρέπει να αναφέρονται στη συσκευασία, να υπάρχει διαφάνεια δηλαδή. Αυτή είναι μια μακρά συζήτηση. Δεν είναι κάτι νέο. Όσον αφορά την κρίση βιοπικιλότητας, και το πώς μπορεί να είναι βιώσιμη η γεωργία ή τι εργαλεία μπορούμε να έχουμε ε, για να μετρήσουμε την ε, βιωσιμότητα διάφορων πρακτικών στη γεωργία, στη χρήση γης κλπ. Εδώ υπάρχουν πολλά εργαλεία και πολλές μέθοδοι. Υπάρχουν. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας. για τις αναλύσεις ροών λοιπά. Είναι τέτοια τα εργαλεία τα οποία μας δείχνουν κατά πόσο κάποιες πρακτικές είναι περισσότερο ή λιγότερο βιώσιμες. Και υπάρχουν και συστήματα πιστοποίησης που έχουν αναπτυχθεί για ένα σωρό είδη. Ε, για την βιωσιμότητα των πηγών και κλπ. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο το θέμα της μέτρησης της βιωσιμότητας, όσο είναι να συμπεριλάβουμε ε, τις παραμέτρους βιωσιμότητας στην πολιτική. Και για τη Γεωργία δεν υπεύθυνη η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, είναι η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Είναι πολύ ισχυρή. Και υπάρχουν και καλά οργανωμένα λόμπι. Ίσως θα πρέπει κανείς να πάει ένα βήμα παραπάνω και να ρωτήσει για τις διαδικασίες ε, βάσει των οποίων εκπονούνται οι διάφορες πολιτικές. Τώρα, ναι, δεν είμαστε πραγματικά μη κυβερνητική οργάνωση. Είμαστε μη κερδοσκοπικοί. Εν πάση περιπτώσει, το ότι δεν κάνει αρκετά Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα λέγω ότι φταίει αυτό καθε αυτό κάποιο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά τώρα είναι προφανές για τον πληθυσμό ότι απαιτούνται ε, περισσότερες και μεγαλύτερες αλλαγές οι οποίες θα επηρεάσουν τον τρόπο ζωής όλων μας. Και ενώ όσον αφορά την ενέργεια η αλλαγή αυτή γίνεται και υπάρχει συνδυτοποίηση και αποδοχή από τον κόσμο, τουλάχιστον στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όχι παντού, πρόκειται για έναν τομέα όπου έχουμε να κάνουμε με δομές, υποδομές, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου χρειάζεται τέτοια αλλαγή. Τα τρόφιμα, για παράδειγμα. Και εξαρτάται η συνέχεια από τις επιλογές του καταναλωτικού κοινού και πάλι είναι δύσκολο πολλές φορές να εξηγήσει κανείς τον κόσμο ε, και να το πείσει ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα για να προστατεύσουμε ε, το κλιματική αλλαγή, να μην γίνεται δηλαδή κλιματική αλλαγή, να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Ε, θα μπορούσαμε ίσως από κοινού με τους πολίτες να συνονεθούμε για το πόσο μπορούν να συμμετέχουν και οι πολίτες περισσότερο σε όλες αυτές τις διαδικασίες μετάβασης και αλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να προχωρήσει πολύ περισσότερο από οικονομικούς παράγοντες που θα πληγούν από τέτοιες πολιτικές. Οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε να χτίσουμε συμμαχίες με τους πολίτες και όχι να βασιζόμαστε μόνο σε αυτούς των οποίων τα, πλεονήματα, τα πλεονεκτήματα πλήττονται. Α, για την άλλη σας ερώτηση, η συνάδελφος θα απαντήσει. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τομείς με τους οποίους θα πρέπει να ασχοληθούμε. Νομίζω ότι ένας σημαντικός τομέας είναι ο οικολογικός σχεδιασμός των προϊόντων και των υλικών συσκευασίας. Θα πρέπει δηλαδή κατά το σχεδιασμό των προϊόντων να σκέφτεται κανείς ε, το τέλος ε, της ε, διάρκειας του προϊόντος. Και στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να αποφεύγουμε αυτό που είπε κάποιος από τους ομιλητές, το να έχουμε τρία διαφορετικά είδη πλαστικών σε, ένα, σε μία συσκευασία, διότι αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα αργότερα κατά την ανακύκλωση. Και μπορεί να μην είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει κανείς τρία διαφορετικά είδη πλαστικού. Να έχει ένα ενιαίο προϊόν συσκευασίας. Αυτό, για παράδειγμα, είναι ένας τομέας που, που με τον οποίο μπορούμε να ασχοληθούμε. Το άλλο είναι ο, ο τρόπος Ε, αποκομιδής των ε, απορριμμάτων ε, πρέπει να μοιράζονται σωστά και πρέπει να λαμβάνουν ε, οι καταναλωτές σωστές πληροφορίες. Υπάρχουν ε, κάποια απορρίμματα τα οποία μπορεί να μαζεύει κανείς ε, ξεχωριστά ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δευτερεύουσα πρώτη ύλη πιο εύκολα. Ο οικολογικός σχεδιασμός η επισήμανση και ο τρόπος ε, ε, συλλογής ε, των απορριμμάτων είναι κάτι που σχετίζεται και με την πληροφόρηση. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε και κάποια άλλα θέματα. Για παράδειγμα, τις μπαταρίες, τους σωρευτές. Έχουμε περισσότερες μπαταρίες από ηλεκτρονικά οχήματα, ηλεκτρικά οχήματα, από ηλεκτρικά ποδήλατα. Όταν παλιώσουν οι μπαταρίες αυτές, θα πρέπει να έχουμε ανακύκλωσή τους στο πλαίσιο της, κυκλική, της κυκλικής οικονομίας. Είναι σχετικά νέο προϊόν αυτό θα πρέπει να βρούμε στρατηγικές για τα διάφορα αυτά προϊόντα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και με αυτό ολοκληρώνεται το δεύτερο σκέλος. Επομένως, συζητήσαμε τις προκλήσεις για το κλίμα, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις υπό την πιο ευρία έννοια, είχαμε και την βιοπικιλότητα και τώρα περνάμε στο τρίτο θέμα ο Νίκολαϊ Πούσκαρεφ ε, για τη δημόσια υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας παρουσιάσει λοιπόν την κατάσταση και τις μελλοντικές προκλήσεις για τις πολιτικές δημόσιας υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αφιερώσω λίγο χρόνο για να σας ε, δώσω μια γενικότερη εικόνα και μια μελέτη για τις ε, πολιτικές δημόσιας υγείας που ε, κατάρτισε το European Public Health Line ακριβώς για αυτή τη συνεδρίαση. Ο βασικός στόχος λοιπόν της μελέτης ήταν να παρουσιάσουμε μια εικόνα των θεμάτων και των ευκαιριών πολιτικής που μπορεί να διαμορφώσουν ε, το θεματολόγιο δημόσιας υγείας της Επιτροπής ΕΜΒΗ για την παρούσα θητεία. Δεν καλύψαμε βασικές πολιτικές για την κλιματική αλλαγή αλλαγή, τις περιβαλλοντικές πολιτικές και την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό μα το είχαν ζητήσει κατά την παραγγελία της μελέτης. Αλλά φυσικά όλα αυτά μπορούν να έχουν πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία. Ε, με επίσης ε, τα θέματα της ποιότητας του αέρα. Ε, κυρίως αποκλειστικά χρησιμοποίησαμε έγγραφα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες και φυσικά τον ΠΟΗ και τον πανεπιστημιακό κλάδο. Το περιεχόμενο με μια ματιά. Καταρχάς, έχουμε κάποιους βασικούς ορισμούς ε, και κάποιες βασικές έννοιες για τη δημόσια υγεία. Στη συνέχεια συζητούμε τις ευρωπαϊκές εξουσίες για να μπορέσει να δράσει σε θέματα υγείας. Βλέπουμε επίσης τι έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, ε, πράγματα τα οποία έχουν ήδη ανατεθεί δηλαδή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και έχουν σαφή αντίκτυπο ή σχέση με την υγεία. Και επίσης η ουσία της έκθεσης ε, βασικές πολιτικές εξελίξεις ε, και προβλέψεις ε, και τα έχουμε κατηγοριοποιήσει με τρεις θεματικές ενότητες, τα συστήματα υγείας, πρόληψη ασθενειών και προώθηση της υγείας και κάποια πράγματα τα οποία είναι οριζόντια. Πριν ε, προχωρήσω, θα ήθελα να σας πω, δώσω κάποια βασικά στοιχεία για να έχουμε ένα πλαίσιο για τη συζήτηση για τη δημόσια υγεία. Όταν εξετάζουμε έρευνες του Ευρωβαρομέτρου, τουλάχιστον ε, για το διάστημα 2017-2019 υπάρχει σαφής ένδειξη ότι η υγεία είναι βασική ανησυχία των Ευρωπαίων ε, επίσης υπάρχει μία σειρά του ΟΣΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχει μία σειρά που λέγεται Health at a Glass, η υγεία με μια ματιά και λέμε ότι 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να αποφύγουν ασθένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν υπάρξει έγκαιρη παροχή θεραπείας. Τώρα, το προσδόκιμο ζωής ε, παρά το γεγονός ότι κάπου έχουν επιβραδυνθεί οι σε κάποιες χώρες, ε, το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πιο υγιή ε, ζωή. Αν δούμε τα στοιχεία της Eurostat, ε, περίπου το 1 τέταρτο ή το 1 πέμπτο της ε, ζωής ε, κάποιου ε, είναι ζωή με κάποια αναπηρία και αυτό φυσικά δείχνει και πάρα πολύ σημαντικές ανισότητες. Κόσμος ο οποίος είναι ευάλωτος σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο έχει και χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής και πολύ χαμηλότερο προσδόκιμο υγιού ζωής. Επίσης, η υγεία είναι το δεύτερο πιο σημαντικό στοιχείο στις δημόσιες δαπάνες των ευρωπαϊκών χωρών. Περίπου το 10% του ΑΕΠ είναι για τα συστήματα υγείας. Ε, το κατά πόσον αυτή είναι πραγματική δεπέν για την υγεία, αν δούμε το ευρύτερο ε, οικονομικό κόστος ε, της κακής υγείας, έχουμε κοινωνική ασφάλιση ή κόστος για τους εργαζομένους και επομένως το ποσοστό αυξάνεται πολύ περισσότερο. Τώρα, οι πολιτικές της δημόσιας υγείας, ε, από ό,τι φαίνεται, προσφέρουν ε, πάρα πολύ ε, καλές μακροπρόθεσμες επιστροφές στην επένδυση. Ε, μία αναθεώρηση υπολόγισε ότι πρόκειται για 14 προς 1, δηλαδή μία μοναδιά επένδυση μπορεί να μας επιστρέψει 14 μονάδες. Όταν συζητούμε λοιπόν πολιτικές για τη δημόσια υγεία, τι εννοούμε ακριβώς. Πολλές φορές υπάρχει μια τάση να συγχέουμε τις πολιτικές για την υγεία με τις πολιτικές ε, για, την, για τις θεραπείες, για τη φροντίδα για την υγεία. Αυτό όμως δεν καλύπτει επακριβώς ε, τι είναι η δημόσια υγεία. Και όπως βλέπουμε στον ορισμό του ΠΟΗ για το τι είναι υγεία, είναι μια κατάσταση πλήρους ε, σωματικής, ε, ψυχικής και κοινωνικής ευημερία και όχι απλώς η απουσία μιας ασθένειας ή μιας νόσου. Ενώ αν δούμε την περιγραφή της δημόσιας υγείας είναι η τέχνη και επιστήμη της πρόληψης των ασθενειών, της παράτασης της ζωής και της πρόθεσης υγείας μέσω των οργανωμένων προσπαθειών της κοινωνίας. Αυτό δείχνει σαφώς ότι έχουμε ένα πολύ ευρύ φάσμα δράσεων. Μπορούμε να μιλήσουμε λοιπόν για πολιτικές για τη δημόσια υγεία οι οποίες ε, στην ουσία προσπαθούν να προσφέρουν τις δυνατότητες ώστε κάποιος να παραμείνει υγιής, να βελτιώσει ε, ε, την ευημερία του και να ε, προλάβει την επιδείνωση της υγείας τους ή την κακή υγεία. Και φυσικά υπάρχει μια προσέγγιση για την υγεία σε όλες τις πολιτικές που είναι μια απάντηση σε αυτή την οριζόντια φύση της χάραξης πολιτικής σε θέματα υγείας και θέλει να εξορθολογήσει την υγεία ε, ώστε να συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις σχετικές ε, διαδικασίες πολιτικής. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορεί να δράσει σε θέματα δημόσιας υγείας αποφασίσαμε να προσθέσουμε αυτή την ενότητα, διότι σε σχέση με αρκετούς άλλους τομείς υγείας, αυτή η ερώτηση δεν είναι τόσο απλή στην απάντησή της ε, σε θέματα δημόσιας υγείας. Και μάλιστα και μια, εν ώψη μιας ενισχυμένης απάντησης από τη νέα ε, Επιτροπή ε, σε αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για νομοθεσία, όπως τόνισε στις πολιτικές κατευθυντήρες γραμμές η μελλοντική Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εξουσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζονται βάσει των Ευρωπαϊκών Συνθήκων. Οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες για την Υγεία ε, καθορίζουν επιμερισμένη αρμοδιότητα για τα κράτη-μέλη Υπάρχουν κοινέ ανησυχία για την ασφάλεια που περιγράφονται περαιτέρω σε κάποιο άλλο άρθρο και υπάρχει και μια ευρύτερη συμπληρωματική αρμοδιότητα για να υπάρχουν αρκετέ υποστηριστικέ δράσει για την ε, πρόληψη τη ε, κακή υγεία και τη βελτίωση τη υγεία. Επίση, ε, το βασικό άρθρο το οποίο ορίζει την αρμοδιότητα για την υγεία είναι το άρθρο 168 και εδώ έχουμε πάρα πολλέ αρμοδιότητε που εκχωρούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προσφέρει πάσας μορφή ε, στήριξη ε, και καλύπτει το πλήρες πεδίο τη δημόσια υγείας. Ε, έχουμε ένα περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εγκρίνει δεσμευτική νομοθεσία και τονίζει ταυτόχρονα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εναρμονίσει την νομοθεσία των κρατών μελών βάσει του άρθρου 168 με εξαίρεση κάποιων κοινών ανησυχιών για την ασφάλεια. Και επίσης τα κράτη-μέλη διατηρούν την αρμοδιότητα να οργανώνουν τα συστήματα υγείας τους. Ε, κάτι όμως που είναι πολύ σημαντικό ε, είναι ότι το άρθρο 168 προσφέρει και το καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να εξασφαλίζει υψηλό ποσοστό προστασία για την υγεία στην εφαρμογή όλων των πολιτικών της, της νομοθεσίας και των δραστηριοτήτων που ουσιαστικά ε, κωδικοποιεί αυτή την προσέγγιση του υγεία στα πάντα. Health in Και επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες σχετικές νομικές βάσεις για να εφαρμόσει ένα θεματολόγιο δημόσιας υγείας. Αυτό που χρησιμοποιείται πιο συχνά είναι το άρθρο 114 για την εσωτερική αγορά. Για παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε για την οδηγία για τα προϊόντα καπνού και άλλους ε, βασικούς ε, ε, νομοθετικούς ε, ε, στόχους. Έχουμε φορολογία, γεωργία, εμπόριο κλπ. στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί. Πάμε τώρα στο ουσιαστικό σκέλος της μελέτης. Εδώ προσπαθήσαμε λίγο να σας παρουσιάσουμε μία εικόνα για τα θέματα και τις ευκαιρίες οι οποίες θα μπορούσαν να ε, βοηθήσουν να διαμορφωθεί το θεματολόγιο για τη δημόσια υγεία της Επιτροπής ΕΜΒΗ στη διάρκεια αυτής της ηττίας. Και θα ήθελα στα επόμενα λεπτά να σας παρουσιάσω μια γρήγορη ματιά για τα όλα τα θέματα που θα μπορούσαν να ε, ανοίξουν ευκαιρίες για να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις για την υγεία σε θεσμικό επίπεδο. Καταρχάς, έχουμε τις βασικές διαδικασίες που είναι στα σκαριά. Ε, το έχετε στην σελίδα επίσης της MV ε, που λέει Health in Progress και έχουμε διάφορες διαδικασίες ε, οι οποίες είναι αρμοδιότητα της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής συγγνώμη, σε διάφορα στάδια, είτε σε προπαρασκευαστικό στάδιο ή και σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου και με τελείως διαφορετικές διαδικασίες ε, υπάρχει συνήθι νομοθετική διαδικασία, εκτελεστικές πράξεις, ε, πράξη κατεξουσιοδότηση, διαδικασία δημοσιονομική κλπ. Επομένως, ε, περιλαμβάνουν την αξιολόγηση τη τεχνολογία για την υγεία, έγκριση τύπου οχημάτων, πολλές διαδικασίες για τα χημικά, η οδηγία για το πόσιμο νερό, η οποία αναφέρθηκε, ο λεγόμενο μηχανισμό πολιτική προστασία, όπου η ΕΜΒΗ είναι η αρμόδια επί της επιτροπή και υπάρχουν και ε, γνωμοδετικές αρμοδιότητες, κοινή γεωργική πολιτική, το ορίζοντας Ευρώπη και πολλές διαδικασίες που αφορούν τον προϋπολογισμό. Μία ακόμα σαφή ένδειξη για το τι μέλη γενέστε είναι στην ε, επιστολή ε, για, που παραδόθηκε στον υποψήφιο επίτροπο για την υγεία. Έχουμε εδώ στη διαφάνεια φάρμακα προσιτά σε τιμή, εφαρμογή του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ε, το e-health και ο χώρος δεδομένων για την ευρωπαϊκή υγεία, ε, μικροβιακή εντοχή, ε, οι ε, επιφυλάξεις στα εμβόλια, το σχέδιο καταπολέμησης του καρκίνου, το, από το χωράφι στο τραπέζι, η στρατηγική για το βιώσιμα τρόφιμα, τα οποία αναφέρθηκαν και θα είναι αρμοδιότητα του Επιτρόπου για την Υγεία, βελτίωση πληροφοριών στους καταναλωτές στα τρόφιμα που περιλαμβάνει πολλά θέματα και την επισήμανση ε, στην, ε, στο πρόσφυγο τμήμα της συσκευασία και πολλά άλλα θέματα και ένα σχέδιο για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες ε, στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο της φιλοδοξίας για μηδενική ρήπανση. Μετά, ευρύτερα, Έχουμε τις έξι προτεραιότητες στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την Μελλοντική Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι πολλές από αυτές τις προτεραιότητες ε, συνδέονται άρρηκτα με τη δημόσια υγεία. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, διότι έχουμε έξι βασικές προτεραιότητες, αυτή, το Green Deal, ε, το η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την υγεία σε θέματα περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, την ποιότητα του αέρα, η φιλοδοξία για μηδενική ρήπανση, ετοιμότητα και απάντηση σε διασυνοριακές απειλές για την υγεία, που πολύ συχνά σχετίζονται και με το κλίμα. Μετά υπάρχει μία δεύτερη σειρά προτεραιοτήτων που αφορούν ε, θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερία. Ε, και εδώ έχουμε μία σειρά από δραστηριότητες που προγραμματίζονται εδώ, που αφορούν και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, στρατηγική για τα φύλλα, ε, πολιτική για τα παιδιά και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια προτεραιότητα για τα ψηφιακά ζητήματα. Η ψηφιακή υγεία εδώ προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για την ε, υλοποίησή τους. Ε, πολλά θέματα φορούν βέβαια ε, ηθικά ζητήματα, προσωπική ζωή και προστασία, ασφάλεια και ε, πρότυπα της υγείας. Μετά έχουμε δεξιότητες, εκπαίδευση και ολοκλήρωση και εδώ έχουμε εκπαίδευση, αθλητισμό, πολιτισμό και υγεία και υπάρχει και ε, ένα νέο σύμφωνο για το, η μετανάστευση και το άσυλο που μπορεί να περιλαμβάνουν και θέματα ε, ένταξης υπηκών τρίτων χωρών που αφορά κυρίως την υγεία των μεταναστών. Η πέμπτη προτεραιότητα μιας ισχυρότερη Ευρώπης στον κόσμο. Εδώ σαφώ υπάρχει μια ευκαιρία να προσπαθήσουμε να έχουμε παγκόσμια πρότυπα για τις ε, συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων για να αντιμετωπίζουν και ανησυχίες για την υγεία και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια υγεία και εν ώψη της εφαρμογής ε, του θεματολογίου των βιώσιμων στόχων ανάπτυξης. Και τέλος, ε, η έκτη προτεραιότητα που αναφέρονται στις ε, πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές είναι η δέσμευση για να αυξηθεί η ακαιρεότητα και να συμπεριλαμβάνονται τα πάντα στη χάραξη πολιτικής. Δεν θα μπορεί κάποιος λοιπόν να προσάψει κάτι στην πολιτική, σε θέματα ηθικής, ευημερία κλπ. Και υπάρχει το άρθρο 5.3 της Σύμβασης του ΠΟΗ για τον έλεγχο του καπνού, που έχει διαδικασίες ε, για να μην υπάρχει ε, αδικαιολόγητη επιρροή από ε, συμφέροντα για τα θέματα αυτά και υπήρξε και μία απόφαση το 2016 που ε, διαπιστώνει ότι δεν είναι πάντα καλά τα πράγματα, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τίθεται και το θέμα του κατάλληλου διαλόγου με τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών στην ε, χάραξη της πολιτικής. Κατόπιν, δεν θα σας τα διαβάσω βέβαια όλα αυτά, ένα άλλο σημείο εισόδου για να δούμε τι προβλέπεται στο θεματολόγιο είναι διάφορες εκθέσεις από τη διαδικασία refit της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάποιες άλλες μελέτες. Ε, οι βασικές υποχρεώσεις λοιπόν υποβολής εξέθρων οι οποίες ήδη κωδικοποιούνται σε κείμενη νομοθεσία. Υπάρχει ένας ενδεικτικός κατάλογος εδώ, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες επ' αυτών στη μελέτη. Αντιστοίχως, το 2020 είναι ε, χρονιά σταθμός και πολλά πράγματα λήγουν το 2020. Αυτό φυσικά ε, σημαίνει ότι ξεκινά και η όλη συζήτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει ανανέωση, παράτωση ή όχι. Για κάποια εξ αυτών έχει ήδη ε, ζητηθεί ανανέωση, ακόμα και από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν και άλλα θέματα στο τραπέζι, τα οποία αφορούν την ε, κείμενη νομοθεσία, όπως για παράδειγμα την ε, οδηγία για τη διασυνοριακή υγεία, κτηνιατρικά φάρμακα και ε, ζωοτροφές ε, με φάρμακα, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται από το 2022, κανονισμός για την κλινική υγεία κλπ. Υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες στη μελέτη, δεν υπάρχει χρόνος τώρα να σας τις πω μία προς μία. Φτάνουμε λοιπόν σε κάποια συμπεράσματα. Νομίζω ότι ένα από τα πορίσματα της μελέτης είναι ότι υπάρχει ευκαιρία προώθησης της δημόσιας υγείας η οποία εδράζεται σε βασικούς ε, τομείς πολιτικής και όχι μόνο αυτούς που αφορούν τα συστήματα υγείας ή την ε, πραγματική ε, υλοποίηση της, ε, των συστημάτων υγείας, αλλά ε, το γεγονός ότι μπορούμε να βασιστούμε σε διάφορες νομικές βάσεις για να επιτύχουμε τα στόχους της ε, δημόσιας πολιτικής για την υγεία και επίσης ε, για τη μελλοντική νομοθετική περίοδο και τις προτεραιότητες ε, που παρουσίασε η Νέα Επιτροπή, έχουμε αρκετά σημεία για την προώθηση της δημόσιας υγείας και σε θέματα τα οποία όμως είναι βασικές προκλήσεις ε, για το θεματολόγιο της υγείας. Υπάρχουν λοιπόν αρκετές ευκαιρίες. Προφανώς, και αυτή είναι και η τελευταία διαφάνεια, όλες αυτές οι ευκαιρίες δεν θα μεταφραστούν ε, σε άμεση ευθύνη της Επιτροπής ΕΜΒΗ ή του Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για την υγεία. Επομένως, εδώ τίθεται και θέμα Διοργανική συνεργασία και συνοχή τη πολιτική και αυτό φυσικά είναι και κάτι το οποίο ε, περιλαμβάνεται σε όλε τι επιστολέ για την αποστολή του κάθε επιτρόπου. Ε, οι υποψήφοι, οι επίτροποι υποτίθεται ότι θα πρέπει να συνομιλούν περισσότερο μεταξύ του και να ακούν ε, ο ένα τι έχει να πει ο άλλο. και επομένως ε, από εκεί και πέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου θα αποφασίσουν σε ποιο βαθμό και για ποιο θέμα θα πρέπει να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, ε, το τονίζω και πάλι. Και τέλος, ε, τρεις τομείς ε, οι οποίοι ίσως πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής και είναι ίσως όχι τόσο σωστά ε, μέσα στις διάφορες προτεραιότητες που εξετάσουμε. Το πρώτο είναι η πρόληψη μη μεταδιδόμενων ασθενειών, που είναι ο βασικός παράγων ε, θανάτων και νόσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι περίπου το 80% της δαπάνης για την υγεία. Υπάρχουν για παράδειγμα το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβολίου για την οικονομία της ευημερία, ε, όπου τονίζουν τη σχέση μεταξύ της πρόληψης των ε, μη ε, μεταδιδόμενων ασθενειών, βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και διαβίου παροχή φροντίδας, ξεκινώντας φυσικά και από την παιδική ηλικία, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα νέα στρατηγικά έγγραφα όλα αυτά. Δεύτερον, όπως είπα και προηγουμένως, άνθρωποι οι οποίοι είναι κοινωνικο-οικονομικά ευάλωτα ε, και είναι δυσανάλογη η επίπτωση για την υγεία τους ε, και επομένως προτείνουμε να υπάρχουν θέματα κοινωνικής ε, δικαιοσύνης. Ίσως ταυτόχρονα θα ήταν ίσως επιθυμητό να σχεδιάσουμε και να παρακολουθούμε αυτές τις πολιτικές βλέποντας και τι αντίκτυπο θα έχουμε σε ανισότητες σε θέματα υγείας. Και τέλος, ένας ε, σημαντικός τομέας είναι το, το θέμα της χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας. Δύο θέματα εδώ πώς ε, οι διάφοροι μηχανισμοί ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μπορούν να ε, συμπεριλάβουν με πιο στρατηγικό τρόπο θέματα για την υγεία. Και το δεύτερο, από το 2021 και μετά, το παρόν πρόγραμμα για την υγεία θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ ε, και θα ήταν λογικό ίσως να εξετάσουμε κατά πόσον θα υπάρχουν και κατάλληλα κονδύλια στον προπολογισμό για τις διάφορες ε, δράσεις που προβλέπονται. Αυτά λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την ε, προσοχή σας. Ήταν μια σύντομη επισκόπηση της μελέτης, υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες στη μελέτη και φυσικά προβλέπω σε ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή λοιπόν ήταν μια επισκόπηση των θεμάτων που θα δούμε στο θεματολόγιο και σας δίνω τώρα το λόγο για ερωτήσεις επάνω στο συγκεκριμένο θέμα, τη δημόσια υγεία. Ο κύριος Πάλμερ. Ευχαριστώ σας, ευχαριστώ πολύ σας, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Και για το συνοδευτικό έγγραφο, το οποίο είναι πολύ πλήρες. Ήταν πολύ χρήσιμη η επισκόπηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δημόσιας υγείας. μία πρώτη παρατήρηση. Εγώ νομίζω ότι μάλλον καταλήγω σε διαφορετικό συμπέρασμα από σας. Μιλήσατε για ευκαιρίες της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου να προωθήσουμε την δημόσια υγεία. Εγώ θέλω ευκαιρίες με την νομοθεσία για να βελτιωθεί η δημόσια υγεία. Αυτή, αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος της, υγεία, της Επιτροπής μας σε, όλα τα θέματα που συζητάμε. Και νομίζω ότι παίζουν πολύ ρόλο οι λέξεις. Έχει διαφορά η προώθηση από τη βελτίωση. Εμείς πρέπει να έχουμε στόχο τη βελτίωση. Μία ερώτηση. Στα συμπεράσματά σας, ε, στην ανάλυση σας, ε, στην ε, επιστολή του νέου επιτρόπου, Θα έχουμε τη δυνατότητα την επόμενη εβδομάδα να έχουμε ακρόαση ακριβώς για το θέμα αυτό. Αλλά όσον αφορά τη διαφορά ανάμεσα στην πρόθεση και τη βελτίωση, εξετάζοντας την επιστολή του Επιτρόπου, νομίζω ότι έχουμε μία τεράστια χαμένη ευκαιρία. Έχουμε έναν κατάλογο για τα ψώνια, δεν υπάρχει ένα, μια γενική φιλοδοξία για βελτίωση της δημόσιας υγείας του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια λίστα, έχουμε τον καρκίνο, έχουμε το, το αλκοόλ, έχουμε τον καπνό. Και Καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε εσείς εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά οι δικές σας παρατηρήσεις νομίζω ότι θα είναι χρήσιμες. Δεν βλέπω να υπάρχει μια γενική φιλοδοξία, να έχουμε ένα γενικό αφήγημα για το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βελτιώσει την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών δεν αναφέρθηκαν καθόλου οι ανισότητες στην υγεία. Δεν αναφέρθηκε καθόλου η βελτίωση της υγείας των ανθρώπων στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και ωραία, ναι, καταλήγουμε στο θέμα των ε, προτεραιοτήτων, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας εμποδίζει από το να είμαστε πιο φιλόδοξοι στο πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες στην υγεία και το πώς θα βελτιώσουμε την υγεία. Είναι θέμα διατύπωσης. Πριν έρθω εδώ στο κοινοβούλιο, πριν κοινοβουλευτής, ε, ήμουνα στην ε, τοπική αρχή υγείας ε, στην περιοχή μου στο Ηνωμένο Βασίλειο και πάντα ε, με δυσαρεστούσε το ότι δεν μιλούσαμε με αρκετή φιλοδοξία και το ίδιο εδώ δεν είμαστε τόσο φιλόδοξοι όσο θα πρέπει να είμαστε. Δεν ξέρω αν έχετε απόψεις για το θέμα αυτό. Αλλά ίσως έτσι σας έδωσα και μια ιδέα για το ποια θα είναι η παρέμβασή μου την επόμενη εβδομάδα. σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ναι, ναι, <laughs> το βλέπουμε. Εν πάση είναι καλή ερώτηση. Και Πράγματι, κάνατε το βήμα προς την ε, πολιτική πλευρά. Η κυρία Βάης, ως ε, ε, πρώην εργαζόμενη στον τομέα της υγείας ε, και ως ε, επιχειρηματίας, γυναίκα επιχειρηματίας. διότι πρέπει να ασχολούμαστε με τα, θέματα ισότητας, Συμφωνώ ότι υπάρχουν δυνατότητες. Έχουμε όμως και το θέμα της επικουρικότητας, διότι υπάρχουν κάποια θέματα που είναι εθνική υποχρέωση, ενώ υπάρχουν και δυνατότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε πιο υγιή Ευρώπη. Προερχόμενοι από το ΕΛΚ και ε, ούσα πλήρες μέλος της Ήτρε θα ήθελα να πω ότι μήπως θα μπορούσαμε να, καλέψουμε, να καλέσουμε την Επιτροπή Ήτρε να μιλήσουμε μαζί της ε, για τις επιστήμες που έχουν στόχο τη βελτίωση της ζωής. Να ασχοληθούμε με τις στρατηγικές για τους γαλάζιους ωκεανούς, ε, το οποίο αφορά και την Επιτροπή Ήτρε, αφορά όμως και την Επιτροπή Ένβη διότι έχει να κάνει με την υγεία και οι δύο επιτροπές αυτές ασχολούνται με την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, την ενεργειακή επάρκεια. Εγώ πάντως από την πείρα μου στον τομέα της υγείας βλέπω ότι η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πολύ πιο φιλόδοξες ε, χώρες από εμάς ε, στα θέματα αυτά και στο πώς στηρίζουν ε, και νομικά και οικονομικά τις καινοτομίες, πώς γίνονται οι δοκιμές νέων φαρμάκων. Και ναι, δεν έχω ερώτηση να θέσω. Ήθελα να προτείνω να καλέσουμε την Επιτροπή Ήτρε να οργανώσουμε ε, μια ημερίδα, κάτι δημιουργικό όπως ε, σήμερα. Ε, διότι είναι πολύ πιθανό ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να βρεθούν σε ένα κενό ανάμεσα στις αρμοδιότητες των δύο επιτροπών και αυτό θα είναι κρίμα. Πρόταση λοιπόν από μένα. Καλή πρόταση θα την σκεφτούμε. Καλό είναι να το πείτε στους συντονιστές σας και στην Ήτρε και στο περιβάλλον, ώστε όταν συζητάμε για την ημέρηση διαδάξη των συντονιστών να υπάρχει αυτή η πρόταση. Θα φροντίσω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όταν μιλούσαμε, λέει η κυρία Μοντσεράτ, για το σύνολο της υγείας, που είναι και ψυχική και σωματική και κοινωνική. Ήμουνα υπουργό υγεία στη χώρα μου, στην Ισπανία. Ε, πιστεύω ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στα εθνικά συστήματα υγείας στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε προχωρήσει πολύ χάρη στους επαγγελματίες του κλάδου, χάρη στην πρόληψη και χάρη βέβαια και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Όμως, ο μεγάλος στόχος της υγείας βρίσκεται μπροστά μας και είναι η πρόληψη. Γιατί έχουμε ένα προσδόκιμο ζωής. Η Ισπανία μετά την Ιαπωνία είναι η δεύτερη στον κόσμο, όπου χάρη στις έρευνες ε, προχωράμε στην εξέταση των ασθενών συνολικά και σίγουρα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο για ένα καλύτερο πρότυπο η πρόληψη πρέπει να αρχίζει από την αρχή, από τη γέννηση, από την παιδική ηλικία μέχρι την ε, γύρανση. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν είναι να λέμε περισσότερα για την ψυχολογική υγεία και την κοινωνική. Κανένας δεν μιλάει για την απομόνωση, ε, για την ε, θλίψη, που στο κάτω-κάτω εξαιτία οικονομικής κρίσης είχαμε πολλά τέτοια προβλήματα έπειτα ε, την ε, έκφραση, τα ψυχοσωματικά ουσιαστικά ε, φαινόμενα που ξεκινάνε από ψυχικές ή από κοινωνικές αδυναμίες και καταλήγουν στην σωματική υγεία πολλές ε, ασθένειες μπορούν να προβληθούν και έχουμε προλάβει πολλές σωματικές ασθένειες, όχι όμως ψυχικές. Ε, το όταν λέμε ότι πρέπει να τρώμε καλά, πρέπει να αναπνέουμε καλά, αυτά έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ε, επίσης, να μην κάνουμε καθιστική ζωή, ε, να μην καπνίζουμε. Όλα αυτά τα λέμε. Δεν μιλάμε όμως για την πρόληψη τη, στην ψυχική υγεία και την κοινωνική απομόνωση. Πρέπει λοιπόν να μην μιλάμε μόνο για την πρόληψη όσον αφορά τη σωματική υγεία, αλλά και την ψυχική και την κοινωνική. Κάπως αναφερθήκατε στις ανισότητες, στα πιο ευάλωτα άτομα και οικονομικά. Ωραία, ακριβώ περί αυτού πρόκειται. Αλλά είναι πολύ σημαντική η πρόληψη και στο ψυχολογικό τομέα και τον κοινωνικό, εκτός από τη σωματική υγεία, να φροντίσουμε και τα άλλα δύο σκέλη που είναι πολύ σημαντικά. Και αυτά μου λείπουν από την παρουσίασή σας και από τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα δηλαδή να προταθούν και αυτοί οι δύο τομείς. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Άλλη ερώτηση. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι από τις τελευταίες σας διαφάνειες, όπου πολύ σωστά ε, μιλάτε για τις ανισότητες στον τομέα της υγείας και λέτε ότι και αυτό θα πρέπει να είναι ένα θέμα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο μέλλον πρέπει να κάνει κάτι θα με ενδιαφέρε να ξέρω τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα των ανισοτήτων απέναντι στην υγεία. Πέρα από όλα τα άλλα λοιπόν που ρώτησαν οι συνάδελφοι, θα ήθελα να μου απαντήσετε και σε αυτό. Παρακαλώ λοιπόν για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ για τις τόσο καλές ερωτήσεις σας. Πρώτη ερώτηση. για την πρόθεση και την βελτίωση. Φυσικά και εγώ δεν θα μιλήσω μόνο σε σχέση με αυτή την ε, μελέτη, η οποία στόχο είχε να εντοπίσει ε, τα θέματα τα οποία θα τεθούν προς εξέταση στο μέλλον. Οπότε, η συνολική φιλοδοξία και η ρητορική, όπως λέτε. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ζήτημα εδώ. Προσπάθησα ακριβώς να εντοπίσω τα κενά και τις αδυναμίες που τελικά έχουν να κάνουν με αυτή την γενική προσέγγιση της πρόληψης και αυτό συνδέεται και με τη δεύτερη ερώτηση. Ότι δεν υπάρχει πραγματική ρητορική δεν είναι κάτι το οποίο φαίνεται να αποτελεί κεντρικό πυλώνα δράσης για την υγεία. Αν το κοιτάξετε στην πράξη, έχω την αίσθηση ότι στις διάφορες προτινόμενες προτεραιότητες θα μπορούσε να προσθεθεί και αυτό, αλλά σίγουρα δεν προωθείται. Θα έπρεπε δηλαδή να αποφεληθούμε από ό,τι ευκαιρίες υπάρχουν. Δεν είναι κάτι το οποίο έτσι προσφέρεται στις διάφορες κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε δει μέχρι τώρα. Οπότε συμφωνώ μαζί σας. Όσο για την πρόταση που κάνετε για συζήτηση, ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα. Για το θέμα της ψυχικής υγείας. Αυτό ήταν ε, επίσης κάτι το οποίο μας έκανε τύπωση και μας. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο τι προβλέπετε για την ψυχική υγεία. Υπάρχουν κάποιες κοινέ δράσεις, υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες που ολοκληρώθηκαν. Αλλά δεν έχω δει κάτι ξεκάθαρο, τουλάχιστον από την Επιτροπή. Και πάλι στο σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου, το Συμβούλιο ζητάει μια στρατηγική για την ψυχική υγεία. Δεν έχει εγκριθεί μεν ακόμα, αλλά υπάρχει σαν επιλογή. Για μας αυτό εγγράφεται και στο γενικότερο πλαίσιο της πρόληψης. Γιατί είναι από τις μη μεταδοτικές ασθένειες. Οπότε παραμένει ο χώρος γι' αυτό. Και για να επανέλθω λίγο στο θέμα της δημόσιας υγείας, είπαμε ότι πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις μέσα στις οποίες ο κόσμος να μπορεί να ζήσει βάσει των επιθυμιών του και των προσδοκιών του. Αναφέρθηκε μια μελέτη για την απόδοση των επενδύσεων. Βλέπουμε ότι η νομοθεσία είναι αυτή που προσφέρει και την καλύτερη απόδοση. Τι να κάνουμε τώρα για τις ανισότητες στην υγεία αυτές οφείλονται σε κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες συνήθως. Αν δηλαδή μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι από φτώχεια μέχρι απομόνωση, διακρίσεις, τότε ήδη έχουμε προχωρήσει αρκετά και στον τομέα της αντιμετώπισης των ανισοτήτων στην υγεία. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες ειδικέ περιπτώσεις όπου θα έπρεπε να προσεχθούν περισσότερο. Να σας πω για κάτι που εγώ δεν το έχω μελετήσει ακόμα επαρκώς, αλλά υπάρχει από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας πρόσφατα μια έκθεση την ανέφερα και στις διαφανίες μου. Α, όχι στο έγγραφό μου, όχι στην παρουσίαση. Λέει τέλος πάντων ότι υπάρχουν πέντε βασικές προϋποθέσεις στην πολιτική όπου μπορούμε να έχουμε ωφέλη υπέρ της υγείας. Και ένας από αυτούς τους τομέας είναι τα συστήματα υγείας που δεν λέω είναι σημαντικό, αλλά είναι ένα. Αλλιώς θα έπρεπε όλους τους παράγοντες που αναφέρονται εκεί να τους ε, φροντίσει κανείς για να έχει πραγματικά καλή υγεία για τον πληθυσμό του. Ευχαριστώ πολύ. Θα το εξετάσουμε. Με αυτό λοιπόν ολοκληρώνεται η σημερινή συνεδρία. Ε, Είδαμε τις μελλοντικέ ε, προκλήσεις πολιτικής για το περιβάλλον, ε, το κλίμα και τη δημόσια υγεία και όπως αναφέρθηκε και στην αρχή και η ασφάλεια των τροφίμων φυσικά είναι στην εντολή μας και θα υπάρχουν και οι προκλήσεις αλλά δεν ήταν θέμα συζήτησης για σήμερα. Προς το παρόν, με αυτό ολοκληρώνουμε και την ημερήσια διάταξη της ε, Επιτροπής με για αυτή την εβδομάδα. Τις επόμενες δύο εβδομάδες έχουμε ακροάσει. Ε, θα είναι εδώ οι συνάδελφοι και θα ακούσουν τους υποψήφιους επιτρόπους. Η πρώτη συνεδρίαση που έχουμε προγραμματίσει είναι για 6 και 7 Νοεμβρίου, αλλά ε, προς ενημέρωση μπορεί να υπάρχει και επιπλέον συνεδρίαση την εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στις 21 Οκτωβρίου ε, του Οκτωβρίου, συγγνώμη, 21 Οκτωβρίου. Ε, θα το δείτε βέβαια, αλλά θα ενημερωθείτε κιόλα. Απλώ σα προειδοποιώ. Με αυτό ολοκληρώνω τη μερίσια διάταξη για αυτή την εβδομάδα. Ε, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.